Okay, people could take their seats now. We are going to start the meeting. So, um, good afternoon everybody and welcome to our meeting. We have Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε, λοιπόν στην Επιτροπή μας. Θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Καταρχάς η ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία. Δεύτερο θέμα, θα μας επισκεφθεί η εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επιστημιστικού προγράμματο για να μα ε, μιλήσει για την καταπολέμηση τη πείνα. Αλλά να διεκπαιρεώσουμε και τα δικά μα πριν ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, να κάνουμε δύο αλλαγέ, ωστόσο. Να σα ανακοινώσω στο σημείο 7 ότι έχουμε ένα πρόσθετο ζήτημα εκτό από τον κύριο Ντεμπράουερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μα μιλήσει για την Ουκρανία θα έχουμε και τον κύριο Παντσέλ Κασουντέλ από το UNCHR που θα μας ε, παρουσιάσει τις θέσεις τους. Στο σημείο 13 επίσης μια αλλαγή όπου δεν θα ψηφίσουμε αύριο για τα ε, μεταλλεύματα αλλά θα ψηφίσουμε το Μάρτιο κατά πάσα πιθανότητα. Θα γίνει συζήτηση όμως για το θέμα αυτό. Αυτό μετά από αίτημα του συντάκτη της νομοδότησης. Θα υπάρξει λοιπόν αλλαγή απόψεων για τα μεταλλεύματα συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Να καλωσορίσω επίση μια ομάδα επισκεπτών του κυρίου Γιάνσεν. Έχετε προσκαλέσει μια ομάδα εδώ στο πίσω μέρο τη αίθουσα. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να απολαύσετε τη σημερινή συνεδρίαση. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών 20 και 22 Ιανουαρίου. Έχετε μπροστά σα τα πρακτικά. Αν έχετε κάποια σχόλια να κάνετε, να ενημερώσετε παρακαλώ την γραμματεία πριν το πέρα τη συνεδρίαση. Αν δεν λάβουμε οποιαδήποτε σχόλια, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί το θέμα. Στο σημείο 3. Το ίδιο ισχύει και για τα πρακτικά τη συνεδρίαση των συντονιστών τη 27η ε, Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε Ένσταση παρακαλώ στη γραμματεία. θα θεωρούνται συγκεκριμένα. Μία μόνο ανακοίνωση να σας κάνω. Σας είπα ότι θα καλωσορίσουμε στην Επιτροπή μας το Παγκόσμιο Πρόγραμμα, το Παγκόσμιο Αντιστοιχικό Πρόγραμμα, την Εκτελεστική Διευθύντρια. Την κυρία Κούζον και τον ε, κύριο Στυλιανίδη, τον Επίτροπο. Αλλά μετά την ανταλλαγή απόψεων στις 5 το απόγευμα, θα ανοίξει και μια έκθεση. Μια φωτογραφική έκθεση. Με εξαιρετικές πραγματικά φωτογραφίες. Η ιδέα ήταν, και αυτό είναι άλλωστε και ο τίτλος της έκθεσης, να πάρουν οι φωτογράφοι φωτογραφίες οικογενειακών γευμάτων από τις πέντε υπήρους. Για να επιστήσουμε την προσοχή μας στο έργο του Παγκόσμιου Επιστηστικού Οργανισμού τον τρίτο όροφο στις 6.30. Αμέσως μετά την ε, συνεδρίασή μας θα ξεκινήσει η έκθεση αυτή. Ελπίζω λοιπόν να τις δείτε όλοι, να περάσετε όλοι από την έκθεση. Στο πάντα της ημερής διαταξής. Ανακοινώσεις της Επιτροπής. Ε, εξ όσων κατάλαβα δεν έχετε ε, ανακοινώσεις να, κάνει, να κάνετε. Πολύ ωραία. Και περνάμε λοιπόν παρά αυτά στην ώρα των ερωτήσεων, όπου υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση τρία διαφορετικά ερωτήματα από πλευρά των συναδέλφων για διαφορετικά ζητήματα. Από εμένα, το ένα ερώτημα του κυρίου Γκερέρο, το δεύτερο, και τη κυρίας Φάουταλα. Το τρίτο ερώτημα. Στο πρώτο ερώτημα, δεν πρόκειται να σας διαβάσω, έχετε τα ερωτήματα του φάκελό σας, αλλά για να γνωρίζουμε η και ο κ. θα απαντήσει νομίζω, να σας πω ότι το θέμα αφορά τα νησιά Σάγκος. Θα γνωρίζετε ενδεχομένως ότι πριν από 50 χρόνια ε, αναγκαστήκαμε από την κρατική κυβέρνηση να μετακομίσουμε, να μετακινηθούμε, γιατί είχε καταστεί αυτό βάση σχετική. Και τώρα το ερώτημα είναι κατά πόσον θα πρέπει να επιτραπεί στον κόσμο αυτό να επανέλθει, να επιστρέψει στα στην πατρίδα του. Η Βρετανική κυβέρνηση αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια σε ό,τι αφορά την επιστροφή του κόσμου στα νησιά αυτά, στις νήσους αυτές. Το θέμα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν ενδεχομένω ε, οι επιστροφές αυτές και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να συνδράμει. Προ τον κύριο Κρέιγ Μακβέιν, λοιπόν, θα δώσω το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. τα νησιά Τσάγκος που είναι έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου υπάγεται στο τμήμα των, της απόφασης για τα υπερπόντια εδάφη του Νοεμβρίου του 2014 και ανήκει και υπάγεται μάλλον στο παράδειγμα 2 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας Ένωσης για τα υπερπόντια εδάφη. Με βάση την σχετική απόφαση τα εδάφια αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, από προγράμματα τη Ένωση βάσει του προπολογισμού τη Ένωση και από κονδύλια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων από του ίδιου πόρου τη. Γνωρίζετε επίση ότι η απόφαση για τα υπερπόντια εδάφη καθορίζει και τι αρχέ κάτω από τι οποίε παρέχεται από την Ένωση χρηματοοικονομική βοήθεια. Σήμερα η Επιτροπή δεν έλαβε κανένα. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει λάβει έτοιμα χρηματοδότηση τη περιοχή αυτή, ούτε έχει υποβληθεί κάποιο α, σχετικό project ή πρόγραμμα. Για την δεύτερη, το δεύτερο τμήμα τη ερώτησή σα, τι επαφέ με τη Βρετανική κυβέρνηση, δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν πιθανέ συζητήσει με τη Βρετανική κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση επανεγκατάσταση ατόμων στα εδάφια αυτά. Ευχαριστώ. Έχω και μία συνέχεια στην ερώτηση. Στο παρελθόν, ο Επίτροπος Πίμπαγκ είχε πει ότι δεν υπήρχε εμπόδιο στην χρηματοδότηση αν υποβληθεί σχετική αίτηση, αλλά θα έπρεπε να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή από την κυβέρνηση τη Βρετανία. Αυτό λέτε κι εσείς. Δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία μαζί σα για το θέμα αυτό. Αυτό δεν μου λέτε. Μάλιστα, αυτό σας λέω. Όπως σας είπα, και βάσει της συνθήκης και της απόφασης ε, είναι επιλέξιμο το νησί αυτό, αλλά πρέπει να γίνει μια αίτηση πρώτα. Ωραία, ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση από τον Ενρίκη Γκερέρο για τις προετοιμασίες για την παγκόσμια διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έγινε μια συνάντηση πριν από δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη σχετικά. Θέλουμε ενημέρωση από την Επιτροπή. η κυρία Γκαρσία Πίρσεν από την Επιτροπή θα απαντήσει και μετά αν θέλει ο κύριος Γκερέρο το λόγο θα τον δώσω. Ευχαριστώ. Το ανθρωπιστικό σύστημα αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σήμερα. Η παγκόσμια διάσκεψη για το θέμα αυτό θα είναι η πρώτη ιστορικά και θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές με στόχο τη δημιουργία πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των διάφορων εμπλεκομένων στον τομέα αυτό ε, ιδίως δε νέων δομών. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής γίνονται μια σειρά διαβουλεύσεων ανά τον κόσμο. Η περιφερειακή διαβούλευση για την Ευρώπη έγινε στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη Βουδαπέστη. Η Επιτροπή ήταν συμπρόεδρος μαζί με την Ουγγαρία και τη Φινλανδία. Στην... Είχε πάνω από 150 συμμετέχοντες, πολύ μεγάλη. Ετοιμάσαμε και ένα ρόλο για είχαμε και συμμετοχή σε υψηλό βαθμό, ήταν ο κ. Στυλιανίδης και άλλοι. Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση αυτή παρουσίασαν μια σειρά ιδεών και παρουσίασαν και συστάσεις λόγω της εμπειρίας αλλά και της πολυπλοκότητας των εμπλεκομένων ήταν δύσκολο να βρούμε συγκεκριμένες προτεραιότητες και να δίνουμε και μια ρεαλιστική ανάλυση των δεσμεύσεων. Ωστόσο, επήλθε συμφωνία για τις βασικές προτεραιότητες που ανακύπτουν, έμφαση, για παράδειγμα, στους ε, πληττόμενους πληθυσμούς, αναγνώριση της βασικής ευθύνης των κυβερνήσεων για την προστασία του πληθυσμού, τη δέσμευση διατήρησης των ανθρωπιστικών αρχών και την επανάληψη του ότι ο, το διεθνέ Αυτοπιστικό Δίκαιο είναι αυτό που θα καθορίζει κατά βάση την αντιμετώπιση των, εμπλε, των εμφύλιων και ε, διεθνικών συγκρούσεων. Υπήρξε επίσης διε, ε, δέσμευση να υπάρξει με περαιτέρω πρόοδο στην ανθρωπιστική ε, αντιμετώπιση και την διαλειτουργικότητα των φορέων. Επίσης αναγνωρίστηκε από τους συμμετέχοντες ότι η επιτυχία της Συνόδου Κορυφής εξαρτάται από όλους τους εμπλεκόμενους. Γι' αυτό και συμφωνήθηκε οι συστάσεις αυτές να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις ούτως ώστε να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση εν και της Συνόδου. Υπήρξε μια σύνοψη των συστάσεων αυτών που παρουσιάστηκε από τους συμπρόεδρους και νομίζω ότι έχει δοθεί και στη γραμματεία της Επιτροπής σας. Τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχει και ένα πλήρες κείμενο των διαβουλεύσεων που θα το στείλουμε και αυτό στην γραμματεία της ΔΕΒΕ. Οι υπόλοιπε περιφερειακές διαβουλεύσεις ολοκληρώνονται με το καλοκαίρι. Πιο σημαντική είναι αυτή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική λόγω των πολλών ε, ανθρωπιστικών κρίσεων εκεί. Και γι' αυτό το λόγο έγινε ε, στην Κωνσταντινούπολη. Στι διαβουλεύσει αυτέ θα είναι παρούσα η Επιτροπή και θα προσπαθήσει να είναι παρούσα και στι υπόλοιπε διαβουλεύσει. Αφού γίνουν όλε οι διαβουλεύσει, θα γίνει και ένα workshop θεματικό το Σεπτέμβριο στη Βόνη και στην Γενέβη τον Οκτώβριο μια παγκόσμια διαβούλευση στην οποία θα προσπαθήσει να είναι παρούσα η Επιτροπή επίσης. Επίσης θα πάμε και σε, άλλα, ε, σε άλλες εκδηλώσεις και διεθνούς ε, χαρακτήρα στην ε, διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και σε εθνικές συνόδους μερικές φορές στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει η Επιτροπή στη διαδικασία αυτή, έχει και την ευθύνη να λάβει θέση και να επηρεάσει την έκβαση της Συνόδου Κορυφής. Πολλοί μάλιστα από τους συμμετέχοντες περιμένουν κάτι τέτοιο από την Επιτροπή. Γι' αυτό θα διαμορφώσουμε θέση, δεν ξέρουμε υπό ποια μορφή ακόμα, αλλά θα στηρίζεται στην εμπειρία και εφαρμογή και διαμόρφωσης πολιτική τη επιτροπή, αλλά και στις ιδέες που παρουσιάζουν άλλοι εμπλεκόμενοι φορεί. Δεν θα είναι μια ξεκάθαρη ε, δεδομένη θέση take it or leave it, αλλά θα είναι ένα πρόγραμμα πολιτικής με όραμα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που ελπίζουμε να λάβουν υπόψη και άλλοι φορεί Σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα γιατί περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στις υπόλοιπες διαβουλεύσεις. Κάποιες από τις προτεραιότητες ωστόσο ανακύπτουν. Π.χ. η ανάγκη να αναδιαμορφωθεί το διεθνές σύστημα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ό,τι φορά την ποσότητα, την μετρησιμότητα και τον αντίκτυπο, την προσαρμογή στο διεθνές σύστημα για να εξασφαλιστούν συνδέσει μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων στην ανθρωπιστική βοήθεια, ούτω ώστε η ανταπόκριση να ταυτίζεται με την ανάλυση των δυνατοτήτων και των κινήνων και την βούληση να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει να δοθούν κίνητα στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και, και την σημασία να βελτιωθούν οι επιεσιακές δυνατότητες της ανθρωπιστικής βοήθειας, η προστασία των αμάχων και των ε, εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό θα είναι βάση περαιτέρω διαλόγου με το Κοινοβούλιο, τα κρατη και τους επιχειρησιακούς εταίρους. Αυτά ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο θέλει να προσθέσει κάτι. Ένα σχόλιο μάλλον, όχι ερώτηση. Πρώτον, ευχαριστώ για τις πολλές πληροφορίες που μας δώσατε, Επιτροπή. Ελπίζουμε να μας στείλετε τα συμπεράσματα και τις εκθέσεις τις οποίες αναφερθήκατε για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα στην Επιτροπή, στην Ανάπτυξης τι θέλετε να κάνετε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό η, να έχουμε μία εικόνα της, ε, των διαβουλεύσεων στην Μέση Ανατολή και την ε, Βόρεια Αφρική Εκεί συγκεντρώνονται δύο από τις πιο σημαντικές κρίση ανθρωπιστικού χαρακτήρα και μέσω και μια τρίτη. Και να σας συγχαρώ διότι η Ευρωπαϊκή Διαβούλευση είχε πολύ εκτεταμένη συμμετοχή και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια συγκέντρωση των προτεραιοτήτων που πηγαίνει προς τη γραμμή που ακολούθησαν κάποιοι από τους στόχους της ανθρωπιστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι στην προετοιμασία της θέσης της Επιτροπής, ε, στην οποία αναφέρθηκε εκπρόσωπος της Επιτροπής, παρότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προτεραιότητες, νομίζω ότι η έμφαση είναι εξίσου σημαντική με τις προτεραιότητες. Τι εννοώ με τον όρο έμφαση. Μια θέση που θα επιτρέπει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν σε ένα κοινό συνεκτικό τρόπο για την προάσπιση του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής που είναι η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο για ανθρωπιστική βοήθεια και που θα γίνει τον επόμενο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω ότι το 2015 θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε από κοινού σε πολλές από τις βασικές συναντήσεις που έχουν και για την αλλαγή του κλίματος και για, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους ε, Ανάπτυξης και τους νέους στόχους της χιλιετίας που θα στη συνάντηση του φθινόπωρο στη ΣΥΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρημα... και στη χρηματοδότηση ανάπτυξης, όλες αυτές οι... όλοι αυτοί οι στόχοι είναι σταθμοί το δρόμο που θα διαμορφώσουν τη θέση της Ένωσης το 2016, συγγνώμη, για να παραμείνουμε όπως είμαστε τώρα ο μεγαλύτερος δρόν σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και σε θέματα ανάπτυξης. Και τα δύο μπορούν να συνδυαστούν μέσω της διαδικασίας link, όπως το λέμε, μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, ούτως ώστε να παράσχουμε και αντοχή, resilience και διάρκεια στη δράση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και μία ερώτηση από την κυρία Χάουταλα. Να σας δώσω το λόγο μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ερώτηση αυτή αφορά τις υποχρεώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε σχέση με το πόσο θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει αυτό το επίπεδο βοήθειας Νομίζω ότι ο κύριος ε, Μακουέιτ θα απαντήσει αυτή την ε, ερώτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρα. Κατρεχάς, παρά το γεγονός ότι έχουμε δημοσιονομικά προβλήματα, τα κράτη-μέλη, ε, φτάσαμε σε ψηλότερο επίπεδο αναπτυξιακή βοήθεια το 2014 1,4% ήταν ε, η αναπτυξιακή βοήθεια το 2013. Μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, ειδικότερα κατά την περίοδο πολύ σημαντικών δημοσιονομικών περιορισμών. Όπως έλεγε η πρόσφατη ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Παγκόσμια Συμφωνία για την Εξάλληψη της Στόχιας, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ισχυρίζεται ότι μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους, τους, ε, τις στόχους της για ε, το ποσοστό της αναπτυξιακής βοήθειας. Εμείς θέλουμε αυτό το ποσοστό να γίνει αποδεκτό από όλες τις χώρες και θέλουμε να ζητήσουμε από όλες τις χώρες να συμμετέχουν στη βοήθεια ανάπτυξης των φτωχότερων χωρών. Πρέπει όμως να υπάρξουν εθνικά σχέδια για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει έκκληση στα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις τις υποχρεώσεις τους και να παρακολουθήσουν τις ε, προόδους τους ε, μέσω της ε, ετήσιας έκθεσης για την παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας. Περιμένουμε για το 2014 την έκθεση, το, τον Απρίλιο του 2015 και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό γιατί κάποια κράτη-μέλη μας είπαν ότι είχαν είχε ακουστεί ότι δεν θα δημοσιευτεί αυτή η έκθεση. Αντιθέτως θα δημοσιευτεί και μάλιστα νωρίτερα Όσον αφορά τώρα ε, την δημοσίευση των ε, αριθμητικών στοιχείων ε, για την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει με ξεχωριστά συμπεράσματα ή ως τμήμα ευρύτερων συμπερασμάτων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ακόμη και αν είναι σημαντική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και είναι καταλήτης της ενίσχυσής μας προς τις χώρες υποανάπτυξη, πρέπει να τα δούμε τα πράγματα σε ένα ευρύτερο στόχο στόχο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και βάσει των στόχων που έχουμε θέσει για μετά το 2015. Πρέπει να δούμε επίση και το πώ μπορούμε να διοχετεύσουμε μέσω και του ιδιωτικού τομέα ε, όλα αυτά τα ποσά και τις, ε, σημα, τις σημαντικές αυτές επενδύσεις. Κυρία Χάταλα, ε, Χάουταλα, μήπως θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, βεβαίως, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη της διεθνούς διάσκεψης ε, ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τις ε, δεσμεύσεις της για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια γιατί ε, το να μην υπάρχουν αυτές οι υποχρεώσεις υπήρχε πάντο, πάντοτε ένα πρόβλημα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις αν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, ε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο απογοητεύει τις ε, χώρες ε, δικαιούχους της βοήθειας Γι' αυτό χαιρετίζω τα όσα άκουσα για την ε, κατάσταση, τον απολογισμό της κατάστασης ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και ξέρω ότι θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για τη χρηματοδότηση ε, της αναπτυξιακής βοήθειας ε, στην περχόμενη σύνοδο που θα αφορά το θέμα αυτό τον Μάρτιο Πρόεδρος, ναι, από ό,τι κατάλαβα θα υπάρξει αυτή η επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει, ε, έχω δίκιο. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ε, για ποιο ακριβώς ε, σημείο ζητάτε επιβεβαίωση, ότι θα συζητηθεί στην Υπουργική ή ότι θα δημοσιευθεί έκθεση. Κυρία Χάουταλα, το δεύτερο, γιατί η πρώτη ερώτηση απαντήθηκε ότι θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δηλαδή. θα δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το 0,7% του ΑΕΠ ε, ανεξαρτήτως του ε, τι άλλοι διεθνείς ε, εταίροι θα πράξουν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Για το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, ε, σαφέστατα ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια έκθεση ε, νωρίτερα βέβαια δεδομένων των συνθηκών αυτής της χρονιάς και η έκθεση θα συμπεριλάβει και κάποια σύντομη ε, ενημέρωση για την χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση των, της εφαρμογής των στόχων, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συζητηθεί το θέμα αυτό από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο, αλλά δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τα αποτέλεσμα των συμπερασμάτων ε, του, ε, και, το, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κατόπιν της ανακοίνωσής μας τη 15 η Φεβρουαρίου. Γνωρίζετε νομίζω την ανακοίνωση αυτή, δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο για την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 0,7, οπότε πρέπει τώρα να πείσουμε τους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο να συμφωνήσουν ε, τουλάχιστον στις 12 Μαρτίου στην ανεπίσημη υπουργική διάσκεψη. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να μιλάμε με τους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε έτσι την ώρα των ερωτήσεων να σας υπενθυμίσω σε όσους είστε νέοι στο Κοινοβούλιο μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις οι οποίες θα εγγραφούν κάποια στιγμή στην ημερήσια διάταξη της ε, Επιτροπής μας ε, τουλάχιστον τρεις μέρες πριν όμως από την, ε, από την συνεδρίασή μας. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε πολύ καλά και βλέπουμε και στις τηλεοπτικές μας οθόνες κάθε βράδυ την ε, ε, εξαθλίωση των ε, ανθρώπων στην Ουκρανία, της πολύ δύσκολες κατάσταση, κατάσταση συνεχίζονται οι συγκρούσεις παρά το γεγονός ότι έγινε κατάπαυση του πυρός, Ελπίζουμε ότι αύριο θα ε, σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Πολλοί ε, είναι αυτοί που υποφέρουν. Η δική μας Επιτροπή είναι υπεύθυνη ε, για ανθρωπιστικά ζητήματα όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο εκτός Ευρώπης, αλλά και εντός Ευρώπης. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε στην ανθρωπιστική αυτή κρίση. Χαίρομαι λοιπόν που στο πλαίσιο αυτό έχουμε εδώ μαζί μας τον Ζων Λουί ε, Ντεμπράουερ, τον ε, Διευθυντή Επιχειρήσεων στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, όπως επίσης και τον κύριο Βενσόν Κοστέλ, ο οποίος είναι ε, Διευθυντής της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ δραστήρια ήδη ε, μέσω του κυρίου Στυλιανίδη, του Επιτρόπου, ο οποίος θα έρθει μάλιστα να μας επισκεφθεί στις 5 η ώρα σήμερα. Έχουμε λοιπόν όλοι ενημερωθεί, γνωρίζουμε την κατάσταση. Το θέμα είναι αν αυτά που κάνουμε είναι αρκετά και τι παραπάνω μπορούμε να γίνουμε. Λοιπόν, να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ντεμπράουερ και ίσως θα μπορούσε να μας περιγράψει την κατάσταση, πώς έχει επιτόπου η ε, βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά ο κύριος Κοστέλ θα μας δώσει μια πιο λεπτομερή περιγραφή για την κατάσταση των ανθρώπων στις ε, ε, περιοχές. Μήπως θα μπορούσατε να περιοριστείτε σε 15 λεπτά. Κύριε δεν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας ξαναδεχθήκατε στην Επιτροπή σας. Θα είμαι σύντομος, το υπόσχομαι. Χαίρο που μπορώ να μετάσχω στην συνάντησή σας ε, σήμερα με πολλούς βουλευτές και με τον συνάδελφο και φίλο Βενσάν Κονστέλ σε ό,τι αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών, ιδίω δε είπε τη αρμοστίας για το θέμα τη Ουκρανίας. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται ε, με εκθετικό τρόπο και εξαιρετικά ανησυχητικό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι αν δούμε τι γινόταν πριν ένα χρόνο και τι προβολές, τι προβλέψεις κάναμε όταν είχε ξεκινήσει ε, η χρήση 2014, κανείς δεν είχε αναφερθεί σε νούμερα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κατάλαβαν σαν βάση της νέας πρόσκλησης ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας θα μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες στη δική του παρουσίαση. Επιτρέψτε μου ωστόσο εισαγωγικά να υπογραμμίσω ότι ο αριθμός των εσωτερικά μετακινηθέντων είναι περίπου ένα εκατομμύριο σήμερα από τα 5,2 εκατομμύρια ατόμων που επιβιώνουν ακόμα στις ε, εμπόλεμες ε, και ε, συγκρουσιακές περιοχές, 3 εκατομμύρια όπως εκτιμάται, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον αριθμό των εμπλεκόμενων ανθρώπων, το, το μέγεθος του πληθυσμού, αποτελεί και μια ποιοτική σχεδόν πρόκληση θα έλεγα, διότι όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προβλήματα, ουσιαστικά προβλήματα προστασίας που εμφανίζονται σήμερα για τον άμαχο πληθυσμό στην περιοχή και βεβαίως υπάρχει μια σειρά προβλημάτων πρόσβασης ε, των ε, εργαζόμενων στα ανθρωπιστικά ζητήματα, πρόβλημα που, γίνεται, όλο και περισσότερο, διότι η ελευθερία κίνησης των ε, εμπλεκομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια περιορίζεται κάθε μέρα. Επίσης, πρέπει να υπογραμμίσουμε το ρόλο που μπορεί να παίξουν ή παίζουν οι αρχές του Κιέβου και η Ουκρανική κυβέρνηση. Ε, αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική βοήθεια προς τους διοχθέντες πληθυσμούς και οι μικρέ τα μικρά κοινωνικά επιδόματα που προβλέπονται είναι περιορισμένα και σε κάθε περίπτωση απειλούνται από την εξάντληση των κρατικών πορών της Ουκρανίας εν γέννη, όχι μόνο ε, για την περιοχή αυτή. Και άλλωστε η κρίση που πλήττει τη χώρα θα είναι μια κρίση που θα ξεπερνά την εμπόλεμη περιοχή, γενικότερα δηλαδή για τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στη χώρα. Η άποψή μας είναι ότι τρεις θα είναι οι στόχοι της να ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάλυψη βραχυπρόθεσμα των άμεσων αναγκών του πληθυσμού, ιδίως ε, σε νερό, ανάγκες μεσοπρόθεσμα των διωγμένων πληθυσμών όταν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις περιοχές προέλευσής τους ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη τόσο κοινωνική όσο και οικονομική και ενίσχυση των ικανοτήτων των Ουκρανικών αρχών. Θα επανέλθω στο ρόλο που πρέπει να παίξει η κυβέρνηση και αρχές της Ουκρανίας, σε κεντρικό επίπεδο τουλάχιστον, για να θα επανέλθω στο ρόλο των τοπικών αρχών, αλλά σαφώς τονίζεται η ανάγκη του ρόλου των κεντρικών αρχών, περιλαμβάνεται και στην επιστολή που, του κύριου Στυλιανίδη που λάβατε κι εσείς, Πρόκειται για ζητήματα που νομίζω ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς η Ουκρανική κυβέρνηση. Όπως είπατε, Πρόεδρε, η Ένωση ήταν δραστήρια εξ αρχής. Η ΕΚΟ έστειλε στο Κίεβο ειδικού στα ανθρωπιστικά από πέρυσι την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014. Γρήγορα δώσαμε και χρηματοδότηση, μικρή στην αρχή, γιατί όπως σας είπα στο ξεκίνημα η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης ήταν τέτοια που δεν μπορούσε κανείς να, προ, να προκαταβάλει να προκαταλάβει συγγνώμη την κατάσταση. Ωστόσο κινητοποιήσαμε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα στη διάθεσή μας μπορώ να επανέλθω σε λεπτομέρειες αυτό αν θέλετε και ενισχύσαμε την ανθρωπιστική μας παρέμβαση ούτως ώστε αφήνοντας τα διάφορα εργαλεία που έχουμε και την συνεισφορά των κρατών μελών το 2014 το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Ουκρανίας στην κατα... της βοήθειας στην Ουκρανία ήταν γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. τα κράτη-μέλη είχαν δώσει 47,5 εκατομμύρια και 32 περίπου η Ένωση. Προπολογισμό της Ένωσης. Εμείς την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια την συμπληρώσαμε με παροχή σε είδο ενεργοποιώντας τον μηχανισμό αλληλεγγύη πολιτικής προστασίας βάσει ενός καταλόγου αναγκών που μα είχε στείλει σε πολλές διαδοχικά μια σειρά κειμένων η Ουκρανική κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι η απάντηση στο τομέα αυτό ήταν λιγότερο δυναμική, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και τις συνεισφορές των κρατών μελών και την ε, δουλειά της Ένωσης. Είχαμε τρία αεροπλάνα κάργο, περίπου ταυτόχρονα με την επίσκεψη του κυρίου Στυλιανίδη. Πρέπει ωστόσο στο θέμα των παραδόσεων σε είδο να είμαστε προσεκτικοί. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που διαθέτει στην ελεύθερη αγορά πολλά από τα είδη πρώτης ανάγκης, δεν χρειάζεται να τα εισάγουμε. Με την ευκαιρία της επίσκεψης του κυρίου Στυλιανίδη αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε αυτό που σε καλά γαλλικά λέμε gap feeding, δηλαδή συμπληρώνοντας τυχόν κενά της εθνικής αγοράς από τη διεθνή αγορά που έπρεπε να παραδοθούν ανάλογα με, την, με, το επίγον, με τον επίγοντα χαρακτήρα. Μέσω ή μακροπρόθεσμα και μετά το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χρειάστηκε να ακολουθήσουμε την πιο αποτελεσματική οδό, να μην παίρνουμε δηλαδή προϊόντα που θα μπορούσαμε να βρούμε στην εσωτερική αγορά. Βρήκαμε ένα τρόπο συνεργασίας ε, προς το παρόν. Πήραμε και κατάλογο ε, αναγκών από την Ουκρανική κυβέρνηση. Λείπουν φάρμακα, ιδίως για κάποιες ιδιαίτερες ασθένειες και λείπει και ιατρικό προσωπικό. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή. Στην συνεργασία με τα κράτη-μέλη ελπίζουμε να μαζέψουμε περισσότερα, να έχουμε περισσότερα μέσα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ την προσοχή στο ότι αυτή τη στιγμή 60 περίπου τα 100 της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται στις περιοχές που βρίσκονται υποκατοχή προτοχή των επαναστατών. Ξέρετε δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω εγώ ότι η ανθρωπιστική βοήθεια ε, στηρίζεται στις αρχές της ανεξαρτησίας, της, ε, της ε, αμεροληψίας και της ουδετερότητας. Πηγαίνει στον πληθυσμό, το πληθυσμό όπου και να βρίσκεται. Όπως σας είπα νωρίτερα βεβαίως η δυνατότητα κυκλοφορίας των ανθρωπιστικών εργαζομένων περιορίζεται αλλά καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να παίξουμε κάποιο ρόλο με αποτελεσματικό τρόπο και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες των ε, πληγέντων των πληττόμενων πληθυσμών και στις περιοχές που τον έλεγχο των επαναστατών. Βεβαίως πολλά περιμένουμε και από την Ουκρανική κυβέρνηση. Υπάρχουν προβλήματα καταχώρησης ε, τα μήτρα τη της κυβέρνησης των ανθρωπιστικών οργανώσεων, υπάρχουν ζητήματα φορολογίας, τελωνιακών δασμών που περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της ανθρώπιστική δράσης. Ο κύριος Στυγιαννίδης μίλησε για το θέμα αυτό με τους συνομιλητές στην επίσκεψή του και ενθαρρύνουμε του ε, εμπλεκόμενου να έρθουν σε επαφή μαζί μα για να μειωθεί η σήμαση το πρόβλημα η απόφαση που λήφθηκε να, να σταματήσουν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ε, στις, ε, στους πληθυσμούς ε, που ζουν σε περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών. Τώρα θα ρωτήσω και την, τον συνάδελφο από την ύπατη αρμοστία που έχει παρουσία εκεί. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει ε, το σύστημα των μένων εθνών να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο των μέτρων αυτό. Για το μέλλον τώρα, το ανοίγει ο κύριο Τηλιανίδη και το επιβεβαιώνω εγώ, στο ξεκίνημα του έτους θα χρειαστεί να παρέμβουμε με 15 εκατομμύρια ευρώ αύξησης του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς έχουμε προβλέψει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχω μια κοινή συνάντηση και με εκπροσώπους του, των επιτόπου του Ηνωμένων Εθνών και με κράτη-μέλη για να συζητήσουμε το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας ή της βοήθειας σε είδος και να δούμε πώς θα πείσουμε και άλλους χρηματοδότες πέραν των πρωτομερών να παρέμβουν στην Ουκρανία δεδομένου του μεγέθους της κρίσης. Προφανώς, όπως συχνά, η πραγματική διακοπή των εχθροπραξιών που αναφέρεται πρόεδρε νωρίτερα θα είχε ως άμεση συνέπεια αυτό συνέπεια να, συνέπεια να προκύψουν νέες ανάγκες είτε γιατί θα μπορούμε να φτάσουμε σε πληθυσμού που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τώρα γιατί θα πρέπει να μπούμε στη δεύτερη φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας την επιστροφή των διωγμένων πληθυσμών στις περιοχές ε, αρχικής εγκατάστασής τους. Ξεπέρασα το 15 λεπτό που μου δώσατε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, είμαι έτοιμος να επανέλθω παντώντας αργότερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Τηρήσατε το χρονικό σας όριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα για να μας πει πως ε, η κατάσταση αξιολογείται από δική σας πλευρά στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση να βρεθώ μαζί σήμερα το απόγευμα εδώ κυρίες και κύριοι. Ήθελα να σας δείξω μια μικρή παρουσίαση PowerPoint, αλλά θα προσπαθήσω να το αφήσω κατά μέρος αυτό για να μην σας μιλήσω τόσο πολύ για το τι κάνουμε εκεί, αλλά για να σας μιλήσω πιο πολύ για τις ελλείψεις που έχουμε στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή σε διάφορα την ανθρωπιστική βοήθεια. Βλέπετε λοιπόν στο γράφημα ότι υπάρχει ε, απεικόνιση των εσωτερικά εκτοπισμένων στην Ουκρανία. Έχει διπλασιαστεί το ποσό αυτό, ο αριθμός αυτός από πέρσι το Δεκέμβριο ένα εκατομμύριο με 420.000 εσωτερικά εκτοπισμένου στην Ουκρανία. Τουλάχιστον αυτό είναι, αυτά είναι στοιχεία του Υπουργείου του σχετικού της Ουκρανίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία είναι εσωτερικά εκτοπισμένα και δεν θέλουν να αντιλαθούν στις αρχές γιατί δεν βλέπουν σε τι θα τους ωφελήσει. Άρα είναι πιο πολλοί πραγματικά εκτοπισμένοι. Κάποιοι μένουν στους συγγενείς, κάποιοι ενδεχομένως να έχουν ε, προβλήματα με τις αρχές και δεν θέλουν λοιπόν να δηλώσουν ε, που βρίσκονται στις σχετικές αρχές. Επίσης έχουμε άνδρες από την Ανατολή που δεν θέλουν να καταχωριστούν όταν πηγαίνουν σε ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές γιατί θεωρούν ότι ενδεχομένως να τους αναγκάσουν να ε, μπουν στο στρατό και να υπηρετήσουν. Ξέρουμε λοιπόν ότι η αριθμοί αυτή το 1.420.000, είναι πολύ χαμηλότερος από τους πραγματικά εκτοπισμένους. Δεν θέλω να σας ε, βομβαρδίσω με στατιστικά στοιχεία, αλλά ένας αριθμός που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι 61% των εκτοπισμένων που έχουν καταχωριστεί δηλαδή ως εσωτερικά εκτοπισμένοι, 61% είναι συνταξιούχοι, άτομα που έχουν φτάσει δηλαδή την ηλικία συνταξιοδότησης. Άρα από πλευράς των αναγκών ε, των ανθρώπων αυτών καταλαβαίνετε πόσο ευάλωτοι είναι. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα για τους πιο πολλούς εξ αυτών. Επίσης, να δούμε τι γίνεται και σε σύγκριση με τους εξωτερικά εκτοπισμένους, δηλαδή τους Ουκρανούς που έχουν αναζητήσει άσυλο σε άλλες χώρες γειτονικέ. Άσυλο ή προσωρινή. Προστασία 670.000 είναι αυτοί οι Ουκρανοί που μένουν δηλαδή σε γειτονικέ χώρε. Είναι μεγάλο ο αριθμό αυτό. Και γι' αυτό στην παρούσα φάση είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για άλλε χώρε. Είναι σημαντικό να ξυπνήσουν, να αντιληφθούν το εύρο τη ανθρωπιστική κρίση. Αν δεν ανταποκριθούμε γρήγορα στι ανάγκε, πολύ λυπάμαι, αλλά προβλέπω ότι πολλοί Ουκρανοί θα επιλέξουν να μετακινηθούν. Άρα η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να ειδωθεί όχι μόνο ως ένα μέτρο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ε, ευάλωτων πληθυσμών, αλλά και σε ένα μέτρο σταθεροποίησης των πληθυσμών. Θα πρέπει οι Ουκρανοί, οι διωγμένοι, να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στη χώρα τους, για να μην αναγκαστούν να μεταναστεύσουν. Στην επόμενη διαφάνεια, δύσκολη στην ανάγνωση ενδεχομένω, αλλά φαίνεται που βρίσκονται οι πιο πολύ εκτοπισμένοι. Βλέπετε λοιπόν ότι η πλειονότητα των ατόμων είναι στις τέσσερις επικράτειες που γειτονεύουν με την Τόμπας. Στις περιφέρειες αυτές, στην Όμπλας, ε, υπάρχει το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο μέρος της ανάγκης. Εκεί εστιάζονται πιο πολλές ανάγκες. Πριν από κάποιους μήνες ε, υποθέταμε ότι είναι τόσο μεγάλη χώρα η Ουκρανία και έχει τόσο μεγάλη μεσαία τάξη και θα είναι μεγάλη η δυνατότητα απορρόφησης αυτών των εκτοπισμένων. Αλλά βλέπουμε μια κάποια κόπηση, κόπωση τώρα. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να νοικιάσει διαμερίσματα σε άτομα που έρχονται από τον Τόμπας, γιατί ξέρουν πολύ απλά ότι δεν έχουν φερεγγιότητα δεν έχουν ε, πρόσβαση πολύ στους λογαριασμούς τους από πέρσι τον Απρίλιο. Πολλοί απλά δεν έχουν χρήματα πλέον. Αντιμετωπίζουν λοιπόν πολλά προβλήματα. Διώκονται από τα σπίτια τους, ε, διώχνονται και δεν έχουν κατάλληλα καταλήματα. Τελευταία διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις ε, περιορισμούς, τα ελλείμματα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς ότι είναι πολύ ευάλωτη η εκεχηρία. Ακόμα και σήμερα δεν γίνεται απόλυτα σεβαστή. Και δεν επηρεάζει μόνο αυτό την ικανότητα των ανθρωπιστικών φορέων να περάσουν τη γραμμή επαφής για τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε δυσκολίες να περάσουμε. Έχουμε 7 checkpoints, σημεία ελέγχου, μερικά από υπό εποπτεία της κυβέρνησης, αλλά όχι δεν αντιμετωπίζουμε τόσο δυσκολίες, αλλά πολλοί από τους μη κυβερνητικού ε, φορείς δεν έχουν την ανάλογη ευκολία. ή αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν περνάνε σε περιοχέ που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Η ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί σημείο ανησυχία. Είναι πολύ αδύναμη η αλυσίδα διαταγών, η λογοδοσία στην πολιτική ηγεσία και γενικά αυτοσχεδιάζουν. Πολλοί κόσμος προσπαθεί να περάσει τις γραμμές, δωροδοκεί, γίνεται κατάσχεση των προϊόντων τους και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες όλο και πιο πολλούς ελέγχους στους πληθυσμούς που προσπαθούν να φύγουν από τις ε, περιοχές που δεν ελέγχονται από τις κυβερνήσεις. Τα γυναικόπαιδα περνάνε και οι ηλικιωμένοι, οι άντρες όχι. Πρέπει να αναγκάζονται να μείνουν στον Τόμπας. Αυτός ο περιορισμός λοιπόν στην ελευθερία μετακίνησης δεν επηρεάζει μόνο την ικανότητα των ανθρωπιστικών φορέων να ανταποκριθούν στις ανάγκες του κόσμου, αλλά και την ίδια την ελευθερία μετακίνηση του κόσμου. Κάναμε μια έρευνα σε 2.000 άτομα στις ε, περιοχές αυτές και διαπιστώσαμε ότι μόνο το ίμιση, το 50% του κόσμου αυτού θα ήθελε να επανέλθει στην, ε, στα σπίτια τους στους τόπους από που ξεκίνησαν, από που ήλθαν. Το πιο ιδανικό θα ήταν ασφαλώς να μπορέσουν να αυτοποδέσουν αυτά τα άτομα το σύντομο των δυνατών. Μιλήσαμε για τον διάφορους τρόπους ε, στρατηγικής ε, ρύθμισης ε, και τα μέτρα που έχει λάβει η Ουκρανική κυβέρνηση από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά και αυτό επηρεάζει κυρίως τις, ε, κοινωνικά, τα κοινωνικά ε, επιδόματα, συντάξεις, ε, επιδόματα οικογενειακά και το καθεξής. Αυτό ουσιαστικά σπρώχνει τον κόσμο να μεταβεί σε περιοχές όπου ελέγχονται από την κυβέρνηση προκειμένου να έχουν τα επιδόματα αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση δεν πληρώνει επιδόματα και συντάξει για παράδειγμα, σε περιοχέ όπου δεν έχει κανένα έλεγχο. Αλλά θα θέλαμε να υπάρχει ένα σύστημα μεταφορά χρημάτων, ρευστού, οπότε να μπορούν οι συνταξιούχοι να μένουν στα σπίτια τους, χωρίς να μεσολαβεί η κυβέρνηση. Δεν θα διατρέξω όλα τα σημεία στην διαφάνεια, αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές ΜΚΟ. Δεν έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Υπάρχει πολύ καλή θέληση, πολύ κινητοποίηση της κοινωνίας. Αυτό σίγουρα είναι ενθαρρυντικό. Αλλά υπάρχουν προβλήματα διακυβέρνηση, διαχείριση. Δεν αποτελεί κάτι καινούργιο αυτό στην Ουκρανία. Από πολλέ απόψει, τα προβλήματα αυτά υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Η ικανότητα λοιπόν τη κυβέρνηση να επιβάλλει πειθαρχία σε επίπεδο Υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκηση, ε, είναι κάτι το πολύ περιπλοκό. Ότι συμφωνείτε στο Κίεβο δεν εφαρμόζονται απαραίτητα στις τοπικές κοινωνίες και αντίστροφα. Άρα, αυτό αποτελεί μια πρόκληση για όλες τις προσπάθειες που γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν σε οι μόρφες διακυβέρνησης να συντονίζονται προκειμένου να επιτρέπουν καλύτερο κεντρικό συντονισμό και από πλευρά τη κυβέρνηση. Ένα άλλο λόγο είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχει πιο πολύ αλληλεγγύη από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών λόγω και της γυπνίασης αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η διμερής ε, αρρωγή δεν συντονίζεται. Για παράδειγμα, κάποιες χώρες αποστέλουν ε, κοντέινερ, εμπορεύματα και Καταρχάς, δεν υπάρχουν ανάγκες για κοντέινερ. Δεν θέλουμε κοντέινερ στην Ουκρανία και γιατί όχι. Γιατί όταν υπάρχουν και καθιστώνται μετά από 20 χρόνια ακόμα εκεί υπάρχουν και στην ε, Βοσνία το είδαμε και στην Γεωργία. Δεν θέλουμε τέτοιου είδους βοηθήματα που θα δημιουργήσουν μια παρατεταμένη κατάσταση. Γιατί για να εγκαταστήσει κανείς ένα κοντέινερ πρέπει να ε, εγκαταστήσει νερό, ηλεκτρικό, ποιος θα πληρώνει τους λογαριασμούς, όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Άρα ζητούμε από τα κράτη πραγματικά να συντονίσουν τις ε, διμερείς μορφές αρρωγής με τις ε, πολυμερείς. Ε. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ουκρανία είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να βρούμε πολλά τοπικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αποστέλουμε τόσο πολλά αντικείμενα για την ανακούφιση της κατάστασης. Οι επόμενοι μήνε θα είναι κρίσιμοι. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα σταματήσει να πληρώνει την πολύ περιορισμένη βοήθεια που παρέχει σε κάποια άτομα σε άτομα που έχουν ειδικέ ανάγκε που έδινε ένα ποσό 50 ευρώ τον μήνα. Θα σταματήσει αυτό γιατί έχουν προβλήματα τα ταμεία τη κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχουν πλέον χρήματα για την χρηματοδότηση αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Είναι σημαντικό η ανθρωπιστική βοήθεια να μην αντικαταστήσει αυτό που κάνει η Ουκρανική κυβέρνηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δουλέψουμε μέσω της ε, Ουκρανικής κυβέρνησης μέσω κοινωνικών προγραμμάτων θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν το δικό τους δυναμικό για να έχουν πρόσβαση στα άτομα στη χώρα. Και είναι πολύ δύσκολο. να αναπτυχθούν οι ικανότητες αυτές. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ρευστό και θεωρώ ότι το πρόγραμμα παροχής ρευστού στην Ουκρανία είναι προφανώς ο πιο αποδοτικός τρόπος βοήθειας των Ουκρανών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Είναι δύσκολο όταν βλέπουμε στη τηλεόραση τι γίνεται και μάλιστα ότι γίνεται τόσο κοντά σε εμά. είναι πάρα πολύ δύσκολο και εμεί το ζούμε αυτό μερικές φορές με σκηνές που βλέπουμε από τη Βόρεια Ιρλανδία. Λέει το BBC ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε να δούμε τόσες ε, σκηνές, όμως έχουμε δει ε, και από την πρώην Ιουγκοσλαβία τέτοιου είδους ε, σκηνές. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο και θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Κύριε Γκερέρο. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοστέλ και τον κύριο Μπρόουερ για τις πληροφορίες που μας έδωσαν σε σχέση με αυτή την κατάσταση που όπως είπαν επιδεινώνεται με εκθετικό τρόπο. Είμαστε ενώπιον μιας κρίσης ε, η οποία για μας είναι άνευ προηγουμένου και έχει άμεσο αντίκτυπο σε 4 εκατομμύρια άτομα και ε, σε εκείνους ε, που ε, έχουν εκτοπιστεί και για εκείνους που πλήττονται άμεσα από αυτήν. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γνωστή για αυτό το θέμα έχει συζητηθεί. Και θα ξανασυζητηθεί βάσει του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η δική μας ε, πολιτική είναι σαφής. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ε, ειρήνευσης και κατάπαυσης του πυρός. μια συμφωνία Μίνσκ 2 έχει εξασφαλιστεί ώστε να γίνει σεβαστό το Μίνσκ 1 και για να μην υπάρξει λόγος ύπαρξης Μίνσκ 3. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν κάποια χαρτιά στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως υπάρχει κάτι που εξαρτάται πολύ περισσότερο από μας και αυτό είναι να υπάρξει μια ανθρωπιστική απάντηση από εμά ενώπιον μιας κατάστασης που συμβαίνει στα σύνορά μας και, στη... και μάλιστα για μια χώρα η οποία ε, γνωρίζει αυτή την κατάσταση γιατί προσπάθησε να ε, συνάψει συμφωνία ε, σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική δέσμευση Εμείς βλέπουμε την επανάληψη όλων όσων έγιναν ε, στη δεκαετία του 90 στα Βαλκάνια ουσιαστικά. Μας έλεγαν ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια που να αξίζει το όνομα αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ανθρωπιστικές δράσεις αλλά δεν ε, είναι συντονισμένες ε, με ε, συγκεκριμένη ανάπτυξη δυνάμεων παρά το γεγονός ότι το είπατε κι εσείς κύριε Ντεμπράουερ, γνωρίζουμε τα τρία επίπεδα δράσης, άμεση, στις ζώνες σύγκρουσης, μετά όσον αφορά τους εκτοπισέντες και μετά μια συνδρομή ευρύτερη ευρύτερου χαρακτήρα. Θα ήθελα και ολοκληρώνω λέγοντας αυτό ότι είναι ένα από τα σημεία για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέμβει σε επίπεδο δηλαδή ανθρωπιστικής κατάστασης. Και νομίζω ότι εφόσον αναφέρθηκε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό είναι ε, ο, η καλύτερη ε, δυνατότητα πίεσης για να υπάρξουν αποτελέσματα Δεν υπάρχει λόγο δηλαδή να στέλνουμε διπλά πράγματα που δεν είναι απαραίτητα και να μην ανταποκρινόμαστε στις, ε, στις ανάγκες, πραγματικές. Πρέπει να ασκηθούν πιέσεις ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου θα υπάρξει μια εντολή που θα δώσει τη δυνατότητα συντονισμού των κρατών μελών στο πλαίσιο τη ανταπόκρισής τους ε, στα, ε, στις τέτοιες καταστάσεις. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, να, ευχαριστώ και τους, να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές μας ε, για αυτά που μας είπαν. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έχει κάνει αξιέπαινες ε, προσπάθειες. Ο Επίτροπος ε, Στυλιανίδης μετέβη στην Ουκρανία και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει να αυξηθεί και το επίπεδο συντονισμού. Είδαμε επίσης, ε, παρά το γεγονός ότι είναι κάπως ε, περιορισμένος, ε, υπάρχουν, υπάρχει ένας αριθμός κρατών μελών τα οποία προσπάθησαν να, παρέχουν, να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Και όπως είπε και ο Ενρίκε προηγουμένως, είναι σημαντικό να δούμε ακόμη καλύτερο συντονισμό στο μέλλον ως προς αυτό το τομέα. Ερώτηση και σχόλιο παράλληλα σε σχέση με αυτό που υπόθηκε για την κούραση, την κόποση που φαίνεται να υπάρχει στο ε, ουκρανικό ε, ζήτημα και επειδή εγώ θυμάμαι την κατάσταση στη δική μου χώρα, μια χώρα ε, 4,5 περίπου εκατομμυρίων ε, κατοίκων και κατάφερε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να απορροφήσει περίπου ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισθέντες. Σε σχέση λοιπόν με την ικανότητα των Ουκρανικών αρχών, με εξέπληξε κάπως η δική σας αξιολόγηση για το πρόβλημα που έχουν δηλαδή με την διαχείριση αυτής της κατάστασης. Λάβαμε επίσης και κάποιες εκθέσεις για τα προβλήματα που έχουν ε, και με το θέμα με την πρόσληψη ε, προσωπικού. Το ερώτημά μου αφορά την αξιολόγηση. Δεν θα μιλήσω για ε, το πώς έχουν τα πράγματα στους, ε, στις Ουκρανικές δυνάμεις, αλλά μιλάω για την ανθρωπιστική βοήθεια ε, και όσους είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση και το χειρισμό όλων αυτών των εσωτερικά εκτοπισέντων. υπάρχει ένα πρόβλημα σχεδόν κατάρρευσης του συστήματος. Πώς το βλέπετε εσείς. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον πράγματι θα υπάρξει εκεχηρία. Υπήρξαν διάφορα σενάρια που ακούστηκαν βέβαια και το, για το τι θα γίνει σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο θετικό. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας ως προς αυτό. Ελπίζω τώρα το μικρόφωνο μου να δουλεύει καλύτερο γιατί οι ε, διερμηνείς δεν άκουγαν καλά. Υπήρχαν παράθυτα, ελπίζω να έχει λυθεί το πρόβλημα. Η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι τώρα καθαρότερη η φωνή σας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μας ε, δώσατε μια γενικότερη εικόνα της ανθρωπιστικής καταστροφής. Είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση και είναι καταστροφικό ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η έκκληση για το συντονισμό και για το συντονισμό της αλληλεγγύης συγκεκριμένα ε, είναι πραγματικά πολύ ε, δικαιολογημένη. Ένα ερώτημα το οποίο με ταλανίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ε, ε, κρίσης αυτής και δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο, σίγουρη ότι είναι, είναι της αρμοδιότητός σας, είναι ε, ποιος έχει τη νομική ευθύνη για την ασφάλεια, τη ζωή, όλες αυτές τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή και προσπαθούν να φύγουν από αυτές τις περιοχές και μιλάω για τους πρόσφυγες. Η Μόσχα τώρα ε, αποστέλει στο Κίεβο το, το λογαριασμό του αερίου ε, που χρησιμοποιούν οι περιοχές αυτές. Αυτό είναι, μια, ε, είναι ένα παράδοξο γιατί τελικά ποιος είναι υπεύθυνο για αυτές τις περιοχές οι ρωσικές ή ουκρανικές αρχές. Εσείς συμμετέχετε σε συζητήσεις για αυτό το θέμα από πλευράς ε, Ουκρανικής κυβέρνησης είναι δικαιολογημένο να λένε ότι δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των ανθρώπων αυτών γιατί πιστεύουν ότι βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και ότι είναι στόχος ρωσικών επιθέσεων. Αν όμως τέτοιου είδους ε, υπόθεση φτάσει σε ένα, ε, στο δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έχετε εσείς πείρα τέτοιου είδους ε, υποθέσεων που υπάρχει παραγνώριση των αναγκών των ανθρώπων που ζουν σε μια τέτοια ζώνη εμπόλεμη, ας την πούμε. Επίσης, οι κοινωνικές ε, μεταφορές έχουν σταματήσει. Κατά τη γνώμη σας, αυτό είναι μία νόμιμη απόφαση. Και κατά δεύτερον, είναι πολιτικός ε, συνετή ε, απόφαση αυτή όταν μιλάμε για ανοικοδόμηση εμπιστοσύνης, δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των ε, διαφόρων μερών. Και κάτι ακόμη, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και το γραφείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest ε, θα, θα ε, οργανώσει μια διάσκεψη σε σχέση με τέτοιου είδους ε, παγωμένες συγκρούσεις και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ακούσουμε αρκετά σε αυτή τη διάσκεψη για να ακούσουμε ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν σε τέτοιου είδους περιοχές και σε σχέση με αυτή την αμφιβολία για το ποιο έχει την εξουσία σε αυτέ τι περιοχέ. Μάλιστα. Ήθελα να σα πω το εξή. Να ακούσουμε άλλο ένα γύρο ερωτήσεων, Ενρίκε, θα πάρει πάλι το λόγο. Ναι. ναι. Να σα πω απλά ότι είναι σχεδόν δεδομένο, θεωρείται δεδομένο, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω ότι ανεξάρτητα από το πολιτικό αποτέλεσμα των συμφωνιών του Μίνσκ, αν θα γίνουν σεβαστέ ή όχι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια και να την αυξήσουμε κιόλα. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε το ένα θέμα με το άλλο. Και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση της Ρωσίας για το θέμα. Τι μορφή συνεργασίας έχετε ή τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε και γενικότερα για το ρόλο που παίζει, δεδομένου μάλλον του ρόλου που παίζει η Ρωσία στην όλη κρίση. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και μετά θα ξανακάνουμε, θα δώσουμε το λόγο. Η Χέιντι, αναφερθήκατε ότι μεταξύ αυτών που ζήτησαν άσυλο σε άλλες χώρες 260.000 περίπου ζήτησαν καθεστώς πρόσφυγα στη Ρωσία. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων αυτών οι Ρώσοι το χρησιμοποιούν ως προπαγάνδα για να δουν δηλαδή πόσοι επιλέγουν να ζητήσουν προστασία στην Ρωσία και να μην μείνουν στη Ρωσία. Τι έχει να πείτε από αυτού. Η Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις αυτές που μας δώσατε. Θα ήθελα καταρχά να διαπιστώσω το εξή. Φαίνεται ότι είναι φαινόμενο τη ανθρωπιστική βοήθεια, ότι πάντα υπάρχουν ασυντόνιστε προσπάθειες από διάφορα κράτη-μέλη και επειδή όλοι έχουμε περιορισμένου πόρους, περιορισμένα χρήματα, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει καλύτερη, καλύτερο συντονισμό σε θέματα ανθρωπιστική βοήθεια. Ίσως θα πρέπει επί της αρχής να το συζητήσουμε αυτό τουλάχιστον μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Μιλήσατε για τις κοινωνικές μεταφορές, ότι έχουν τερματιστεί και ότι πάνω από 60% των προσφύγων είναι συνταξιούχοι. Ουσιαστικά μετακινούνται για να πάρουν τη σύνταξή τους οι άνθρωποι. και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό. Να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε να μπορέσει να μείνει εκεί που μένει, να μην χρειαστεί δηλαδή να φύγει, να ενταχθεί κάπου αλλού. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε και δεν έχει ξεκαθαρίσει στο κεφάλι μου είναι πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αν δεν υπάρχει αρκετή διαχειριστική βοήθεια από πλευρά Κιέβου, τι δυνατότητε έχουμε να ασκήσουμε επιρροή και στο Κίεβο προκειμένου να μας δώσει αυτή την διοικητική, διαχειριστική βοήθεια. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό προκειμένου ο κόσμος να πάρει τα επιδοτήματα, τα, χρήματα αυτά. Είπατε ότι είναι μικρά τα ποσά αυτά, αλλά ίσως και γι' αυτό είναι πιο σημαντικό να τα λαμβάνουν ακριβώς τα επιδόματα αυτά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος να προσθέσω κι εγώ κάποια σημεία. Μου φαίνεται ότι είναι κρίμα. Κρίμα να μην συντονίζουν τις προσπάθειες στα κάτι μελη Αναρωτιέμαι κύριε Κώστα μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Έγινε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από λίγο. Τέθηκε το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συντονίσει τα κάτι μελη Και αν ναι, πώς ε, το UNCHR επικοινωνεί με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξηγήσει ότι ε, δεν θέλουμε, σας παρακαλούμε για παράδειγμα, τέτοια αγαθά, δεν θέλουμε κοντέινερ. Μη μας θέλετε προϊόντα εκτός Ουκρανίας, προτιμούμε να τα αγοράζουμε στην Ουκρανία. Με ποιον επικοινωνείτε για τέτοια ζητήματα και τι συμβαίνει με τις πληροφορίες αυτές, ποιος λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές και τι τις κάνει. Υπάρχει κάποιος δανεισμός μεταξύ κρατών μελών, για τον έπολα για παράδειγμα. Αποφασίσαμε να υπάρξει συντονιστικός μηχανισμός, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όχι μόνο της ευρωπαϊκής βοήθειας, αλλά και των ευρωπαϊκών εισαγωγών. Αν ρωτιέμαι μήπω σε τέτοιε περιπτώσει μεγάλων κρίσεων χρειάζεται αυτόματα καλύτερο συντονισμό. Μήπω θα πρέπει να είναι αυτό ένα η αυτόματη αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων. τα ζητά κανείς άλλο το λόγο. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Ο κ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους βουλευτές που έφεσαν τα ερωτήματά τους. Σημαντικά είναι όλα, αλλά πολλά από τα ερωτήματα δείχνουν ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να σεβαστούμε τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής προστασίας σε ένα πολύ πολιτικό πλαίσιο. Εμείς μας τέθηκε ε, μας ερωτήματα για τη θέση της Ρωσίας, για παράδειγμα. Βλέπετε ότι όλη η ατζέντα έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αλλά εμεί πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή να φτάσουμε στους ευάλωτου πληθυσμού όπου μπορούν, όπου έχουν ανάγκη, με επίγνωση, και εδώ απαντώ στην κυρία Χαουταλά, ότι ο κύριος υπεύθυνο τη προστασία των πολιτών παραμένει το Ουκρανικό κράτος. Από όσο γνωρίζω τα πίμαχα εδάφη δεν έχουν αποσπαστεί από το Ουκρανικό κράτος. Η βασική λοιπόν αρχή είναι η αρχή της ευθύνης του κράτους της Ουκρανίας. Ο συνάδελφος εξήγησε ωστόσο πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια λυσίδα ηγεσία ούτω ώστε να υπάρχει ουσιαστική εφαρμογή των αποφάσεων επιτόπου δεν σας είπα στην πρώτη παρέμβασή μου ότι και εμείς προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση της ικανότητας αυτής. Στείλαμε ε, ομάδες ειδικών, όχι ειδικών ανθρωπιστικής προστασίας, αλλά πολιτικής προστασίας για να δημιουργήσουμε εθνικά σχέδια αντίδρασης. Η εντύπωση που έχουν είναι ότι έχουν, έχει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά. Είπατε πρόεδρε και με εντυπωσίασε ότι είναι εκπληκτικό. Δύσκολο μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι δύσκολο να κάνεις ανθρωπιστική βοήθεια σε μια πόλη που είναι αδερφοποιημένη με μια πόλη που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Ε, πρέπει να σας πω ότι όταν βλέπετε εκπρόσωπους των, των Ηνωμένων Εθνών ή των, των ΜΚΟ ε, που έχουν δουλέψει σε χώρε όπω το Καμερούν, το Τσάτ, το Μαλί και προσπαθεί να του εξηγήσετε ότι ίσω η δυνατότητα παρέμβασή σα στι χώρε εκείνε, στη χώρα αυτή πρέπει να περιορίζεται διότι πρέπει να κρατήσετε κονδύλια για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, πραγματικά εκπλήσονται. Εκπλήσονται. Άρα ε, απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμός. Δεν έγινε απόλυτα και θα συμφωνήσω με τα παραδείγματα που ανέφερε ο συνάδελφος Κοστέλ. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους πρόεδρε. Δηλαδή συχνά κάποια κράτη-μέλη, τα γειτονικά κυρίω, θέλουν να δείξουν ότι είναι εκεί, δίπλα. Και άρα το να χρησιμοποιηθεί ένας ευρωπαϊκός συντονισμός είναι μια διοικητική αλλά και πολιτική ε, παρέκβαση. Είπατε, πρόεδρε, από το μυαλό μου το πήρατε, την ανάγκη συντονισμού, μάλλον το συντονισμό που κάναμε για το έμπολα. Ε, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση με τα κράτη-μέλη και θα αναφερθούμε στα κράτη-μέλη την ανάγκη να υπάρξει ένας ε, μηχανισμός συντονισμού για την Ουκρανία παρόμοιος με αυτό του έμπολα. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία με την Ουκρανική κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την αντικειμενική αδυναμία απάντησή της ως μία απάντηση. Επίσης πρέπει να πούμε, και μπαίνω σε έναν χώρο που δεν είναι δικός μου, ότι για μακρύ χρονικό διάστημα η κυβέρνηση της Ουκρανίας για λόγους ε, που μπορεί να, κατα... να κατανοήσουμε, αρνιόταν να δεχθεί τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Εγώ προσωπικά πήγα για πρώτη φορά στην Ουκρανία το καλοκαίρι πριν την έκτακτο, το έκτακτο συμβούλιο του Αυγούστου και εκεί για πρώτη φορά σε κυβερνητικό επίπεδο δέχθηκαν εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της κρίσης ότι πληρούνταν δηλαδή όλοι οι και όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις. Αυτό εξηγεί και την άρρη καθυστέρηση της απάντησης της ουκανικής κυβέρνησης στο ζήτημα. Η χώρα θεωρούσε ότι ήταν μια χώρα ε, σε πόλεμο με αντάρτες εξού και και επανέρχομαι σε αυτό που ρώτησε η κυρία Χάουταλα, εξού και η διακοπή των χρηματοοικονομικών μεταβιβάσεων προ τι ε, περιοχέ υπό τον έλεγχο των ανταρτών, έστω και αν όπω έλεγε ο Βενσάν Κοστέλ σε κάποια μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική αυτή τη απόφαση. σίγουρα η απόφαση αυτή ωστόσο θα έχει ε, καταστρεπτικές, απόλυτα καταστρεπτικές επιπτώσεις στην ε, ζωή και την ευημερία, εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, του ενδιαφερόμενου πληθυσμού. Δεν είναι απόφαση σκόπιμη ε, για την υποστήριξη του πληθυσμού αυτού που όπως ε, σας είπα ε, παραμένουν ακόμα πολίτες της Ουκρανίας μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Άρα το Ουκρανικό κράτος είναι υπεύθυνο για την προστασία τους. Ευχαριστώ. Κύριος Κοστέλ. Εν συντομία, να απαντήσει στα διάφορα ερωτήματα. καταρχά. δεν θα ήθελα να φύγετε από την αίθουσα εδώ, πιστεύοντα ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Φυσικά υπάρχει στρατηγική ανταπόκριση, σχέδιο το οποίο έχει καταστρωθεί από τι διάφορε υπηρεσίε του ΟΗΕ σε συνεργασία με τι ΜΚΟ, σε συνεργασία με του δωρητέ, έχει συζητηθεί με διάφορε χώρε για να διευκολυνθεί και η οργάνωση με την ότσα με το ανάλογη υπηρεσία του ΟΗΕ. Αυτό γίνεται στο Κίεβο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα κόμβο και άλλες ε, σειρές ε, φορτηγών που καταφτάνουν κάπως σπασμωδικά, χωρίς συντονισμός. Πριν από, κάποιες χρόνιες, πριν από κάποια χρόνια διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είπαν ε, από πλευρά του ΟΗΕ εντάχθηκαν να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό, να υπάρχει και αποστολή συγκεκριμένων ομάδων. Και από πλευρά ΟΗΕ έχουμε δύο κλάστερ σε ό,τι αφορά τα καταλήμματα. Υπάρχουν λοιπόν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν βοήθεια διμερός. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει συντονισμός, να σας πούμε τι είδους καταλήμματα χρειάζονται. Τέτοιου είδους ε, συντονισμός δεν υπάρχει ακόμα. Το ΕΚΟ, αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ, προσπάθει να βοηθήσει. Σταδιακά όμως γίνονται όλα αυτά. Μιλήσατε για τα σχέδια της υπηρεσίας ΕΚΟ για να ανταποκριθεί στην κρίση. Η στρατηγική ανταπόκριση του ΟΗΕ ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές είναι οι άμεσες ανάγκες. Δεν περιλαμβάνουν του ενοικοδόμηση των καταστραμμένων τμήματων της χώρας. Είναι σαφές ήδη ότι ο ανθρωπιστικός προϋπολογισμός της ε, Επιτροπής και των κρατών μελών δεν ακούν για να καλυφθούν κάποιες από τις ανάγκες αυτές, κοιτώντας ε, και την πολλαπλασιασμό άλλων κρίσεων που δεν έχουν επιληθεί. Θα πρέπει να ζητήσουμε και άλλου προπολογισμού και άλλη χρηματοδότηση. Και δυστυχώ δεν υπάρχει άλλο τρόπο παρά να κοιτάξουμε και τον προπολογισμό, τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία Ανθρωπιστική Βοήθεια των κρατών μελών. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τη σταθεροποίηση. Υπάρχει πολιτική απάντηση σε αυτό. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρεια. Αλλά στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο οι αρχές που ελέγχουν μια επικράτεια είναι υπόλογε και υπεύθυνε για την προστασία των πολιτών, ακόμα και αν δεν έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη. Στην Υπερπνησσαρία, στην Νότια Σουτία, στην Αυχαζία, στον Αγκόρνα Βραμπάχ, Αυτό λέμε ότι οι αρχέ που ελέγχουν την ε, επικράτεια έχουν και υποχρεώσει έναντι των πολιτών. Αυτό δεν ε, απαλλάσσει λοιπόν τις ε, Ικρανικές αρχές από τις ευθύνες έναντι των πολιτών που ζουν σε περιοχές που, που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, αλλά όπως και να το κάνουμε, οι ευθύνε τους είναι πιο περιορισμένες εκεί. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σήμερα. Οι Ουκρανοί κατά πόσο αναζητούν άσυλο στην Ρωσία. Ναι, και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε παρουσία και στην Ρωσική Ομοσπονδία και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί. Παρέχεται βοήθεια λοιπόν στους Ουκρανούς που καταφθάνουν στην Ρωσία. Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων αυτών δεν βρίσκεται σε μαζικά καταλήμματα, μόνο 30.000. Οι πιο πολλοί μένουν στα συγγενείς τους. Πολλοί Ουκρανοί πάνε λοιπόν στη Ρωσία, αλλά δεν το κάνουν αυτό για ιδεολογικούς σκοπούς. Απλά έχουν ένα συγγενή. Έχουν μια δουλειά που τους περιμένει. Ή επειδή τους αναλαμβάνει η Ουκρανική κυβέρνηση, η Ρωσική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις συντάξεις τους. Το ίδιο και στη Λευκορωσία. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά βλέπουμε και κάποια άτομα να επιστρέφουν από τη Ρωσία στην Ουκρανία και δεν πάνε πάντα εκεί που μέναν σε κάποιες περιπτώσεις πηγαίνουν και σε περιοχές ελεγχόμενες από την κυβέρνηση. Το οποίο καταδεικνύει ότι δεν ήταν ιδεολογικοί οι λόγοι που τους έστειλαν προς την Ανατολή. Απλά είχαν φίλους συγκινείς. Για το θέμα των κοινωνικών επιδομάτων. Το Μάρτι και τον Απρίλιο του περσινού έτους η Ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει την παροχή συντάξεων, μισθών για δασκάλους, νοσοκόμους, γιατί πολύ απλά κατάλαβαν ότι τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν απαραίτητα στον κόσμο. Έχουν ανησυχίες και δηλώνουν ότι δεν θέλουμε να δίνουμε χρήματα που ουσιαστικά τα καταχρούνται οι de facto αρχές στον Τόμπας. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός μηχανισμός που τα χρήματα δεν θα περνάνε από τις συναλλακτικές αρχές της αρχέ. Αυτό είναι δύσκολο ασφαλώ, γιατί δεν μπορεί κανεί να μεταφέρει ρευστό στις γραμμές, ε, πέρα από τι γραμμέ ελέγχου. γιατί φυσικά μιλάμε για τους συνταξιούχους που δεν πρέπει να αναγκαστούν να φύγουν από τα σπίτια τους για να πάρουν την συνταξή τους. Στην πρόσφατη συμφωνία του Μίνσκ στις 12 Φεβρουαρίου υπάρχει μία ολόκληρη παράγραφος που μεταξύ άλλων αναφέρει και τα κοινωνικά επιδόματα. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με αυτό. Υπάρχει και μία παράγραφος με περίεργη διατύπωση σε ό,τι αφορά την ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτούς που έχουν πιο πολλές ανάγκες. Στο τέλος του παράγραφου λοιπόν υπάρχει κάτι το περίεργο. Αναφέρεται ότι Αυτά θα πρέπει να γίνουν βάση διεθνών μηχανισμών. Δεν είμαι σίγουρος τι εννοεί η παράγραφος αυτή γιατί δεν ξέρω τι υπάρχει. Δεν ξέρω και από πού προήλθε αυτή η διατύπωση τελευταία στιγμή. Και βλέπω ότι στον τύπο στη Ρωσία γίνεται μεγάλος λόγος στον τύπο για τους μηχανισμούς αυτούς που θα πρέπει να δημιουργηθούν. Με μεγάλη προσοχή και σοφροσύνη θα πρέπει να, κινηθούμε Προ την κατεύθυνση αυτή, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχουν διαμεσολαβητέ και να υπάρχει πιθανότητα κατάχρηση τη Ευρωπαϊκή βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο σας ε, που ήσασταν εδώ και που ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινείς μαζί μας για τα προβλήματα που υπάρχουν πραγματικά επί τόπου και για τη δύσκολη πολιτική κατάσταση. Πρέπει να προβληματιστούμε νομίζω και εμείς για το πώς ε, θα γίνει ο συντονισμός της ενίσχυσης εντός ε, της Ένωσης και σκέφτομαι αυτά που είπε ο κύριος Γκερέρο να υπάρχει μια συστηματική, ένα συστηματικό συντονισμός της βοήθειας από την αρχή της κρίσης. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε και με τον Επίτροπο ε, τώρα σε λίγο για το πώς μπορεί να είναι πιο αποδοτική αυτή η ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Um, we can't start the next part of our... Δεν μπορούμε να αρχίσουμε πριν από τις 5 το επόμενο σημείο της ημερήσιας διαταξή μας. Ε, ε, γιατί τότε θα έρθει ε, η εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος και ο Χρήστος Τηλιανίδης. Παρακαλώ λοιπόν να διακόψουμε ως τις 5. Σας παρακαλώ να είστε παρόντες γιατί θα έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση ε, με τους δύο προσκεκλημένους μας για το, επιστημιστικό μας, για το, για το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα και την ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων. Παρακαλώ το προσωπικό των ομάδων να αποστείλει email, ε, να υπενθυμίσει στους συναδέλφους μας να είναι εδώ στις 5. Ευχαριστώ. we can Okay, colleagues, we're going to... Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε την συνεδρίασή μας. Χαίρομαι όλος ιδιαιτέρως που είναι εδώ μαζί μας σήμερα η Ερθαρίν Κάζεν, εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος, που ήρθε από τη Νέα Υόρκη, ταξίδευε όλο το βράδυ και το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ένα μισοπαγωμένο τσάι. Είναι εδώ βεβαίως και ο Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, ο Χρήστος Τηλιανίδης. Όσοι ήσασταν και προηγουμένω στην Επιτροπή μας θα γνωρίζετε ότι η κυρία Καζίν δεν έρχεται για πρώτη φορά εδώ. Ήταν εδώ και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ε, θητεία. Και επειδή το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα είναι ένα εταίρος μας στην προσπάθεια καταπολέμησης της πείνας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί συνεργαστήκατε μαζί μας ε, Χαιρόμαστε όλους ιδιαίτερους που είστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Στις 6.30 ώρα θα πάμε και θα εγγενιάσουμε την ε, έκθεση φωτογραφίας ε, για το επιστημιστικό πρόγραμμα για να ευαισθητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί η Επιτροπή μας είναι μικρή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να γνωρίζουν το πρόγραμμα αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση ε, από απόψε ως ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στους δύσκολους καιρούς μας. Υπάρχουν πολλές κρίσεις ε, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Αφρική. Μόλις μιλήσαμε και για την Ουκρανία. Μίλησα για, με την κυρία Κάζεν για το, το πώς συνεισφέρει το Παγκόσμιο Επιτιστικό Πρόγραμμα στην Ουκρανία. Επίτροπε Στυλιανίδη, γνωρίζω ότι δεν έχετε ανασάνει από τη στιγμή που αναλάβατε το, το χαρτοφυλάκια σας. Ε, ε, είχαμε το θέμα του έμπολα, είχαμε το θέμα της ε, διόρυγας της Γάζας, είχαμε το θέμα του Μαλή. Είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψηφίσματά του πρόσφατα έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους ε, πλήττονται στο Ιράκ και τη Συρία. Μόλις ε, ε, εγκρίναμε και ψήφισμα για την Ουκρανία και εγκρίναμε και ένα ψήφισμα για την παιδική κακή διατροφή. Νομίζω ότι ήσασταν παρόν. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ δραστήριοι για τα θέματα αυτά. Του χρόνου έχουμε και την Παγκόσμια Σύνοδο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζετε ότι έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς, έχουμε προκλήσεις και από δημοσιονομικής απόψεως. Πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Το συζητήσαμε και για το θέμα της Ουκρανίας. Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού εντός της Ένωσης. Πολλά λοιπόν πρέπει να γίνουν. Και γι' αυτό χαίρομαι όλος ιδιαίτερω ε, που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα επίση να σημειώσω, το Σεπτέμβριο θα γίνει και η σύνοδος του ΟΗΕ για ε, τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Θέλουμε μηδενική πείνα, αυτό είναι ο στόχος μας. Ε, έχουμε και τον ε, εισηγητή μα για το θέμα αυτό και άλλους συγητές σχετικούς με το θέμα αυτό το, να, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και δεν έχουμε ακόμη ε, επιτύχει βασικούς στόχους της χιλιετίας, υπάρχουν ε, παιδιά τα οποία όχι μόνο υποσυτίζονται, αλλά δεν, δεν μπορούν καθόλου να τραφούν. Ε, πρέπει τουλάχιστον να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της πείνας σε περιοχές όπου συμβαίνουν ακόμη τέτοια πράγματα στον 21ο αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να δώσω το λόγο στην κυρία Έρθαριν Κάζεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Επίτροπε, με τη Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για να που ανταλλάσσουμε και πάλι απόψει σε θέματα ανάπτυξη μαζί με τον Επίτροπο Στυλιανίδη. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την δεύτερη αυτή ευκαιρία που μου δίνετε να εμφανιστώ εδώ στην Επιτροπή σα. Επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω τη σημασία του έργου σας καταρχάς που είναι κρίσιμο για να μπορέσει να διατηρηθεί το θέμα του, ε, της σωστής διατροφής, της επαρκούς παροχής ε, τροφίμων στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, των παγκόσμιων, ε, και της παγκόσμιας ατζέντας. Άλλο θέμα να συζητάμε θέματα χρόνιου υποστατισμού και άλλο πράγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή σας να αναγνωρίζει ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί σε όλες τι πλευρές του κόσμου. Οι συζητήσει σα και οι δικέ σα αποφάσεις δημιουργούν την πολιτική βούληση που χρειαζόμαστε απαραίτητο στον τομέα για να βοηθήσουμε όλους εκείνους όσοι προσπαθούν να έχουν τρόφιμα για τις οικογένειάς τους και που θέλουν τις βοηθήσεις να βγουν από το καθεστώς του υποσυντισμού για να πετύχουμε ένα κόσμο χωρίς καθόλου πείνα, με μηδενική ανοχή στην πείνα σε βιώσιμο επίπεδο. Από το 2013 όταν παρουσιάστηκα για τελευταία φορά εδώ στην Επιτροπή σας έχει ξεσπάσει τεράστια κρίση σε όλο τον κόσμο, κυρία Πρόεδρε, Και παρά το γεγονό ότι η διεθνή κοινότητα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο για να μειώσει τον αριθμό ατόμων που υποφέρουν από πείνα. Στα 850 εκατομμύρια, 805 εκατομμύρια, η σκληρή αλήθεια είναι ότι ποτέ πριν δεν είχαν απαιτήσει τόσο πολλά οι κρίσει από τι ανθρωπιστικέ οργανώσει. Έχουμε πιο πολλού πρόσφυγε ουσιαστικά από ό,τι είχαμε από τον παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Και αυτή η κρίση, αυτές οι κρίσει, θα ήταν τεράστιε απαιτήσει και στο δικό μα το πρόγραμμα, στο παγκόσμιο επιστημικό πρόγραμμα. Χρειάζονται λοιπόν όλο και πιο πολλοί βοήθεια για παροχή τροφίμων, γιατί πολύ συχνά δεν χρειάζονται μόνο τρόφιμα. Αναγνωρίζεται πλέον ότι σε πολλά μέρη υπάρχουν τρόφιμα. Η πρόκληση είναι η πρόσβαση στα τρόφιμα αυτά. Υπάρχουν τρόφιμα, αλλά οι φτωχοί και οι ευάλωτοι αυτοί που ε, έχουν πληχθεί από τις αρρώστιες όπως ο εμπόλα ή τον πόλεμο όπως η Συρία δεν έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα αυτά. Άρα, χρειάζονται εργαλεία προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε τα τρόφιμα αυτά. Είτε πρόκειται για ρευστά χρήματα, είτε πρόκειται για βάουτσερ, είτε πρόκειται για βοήθεια οργανωτικής φύσεως. Είτε πρόκειται για βοήθεια από αέρος το πρόγραμμα, το Παγκόσμιο Επιστημικό Πρόγραμμα και οι εταίροι μας ανταποκρινόμαστε και σε αυτές τις ανάγκε. Αναγνωρίζουμε το τι χρειάζεται ο κόσμος και όχι τι θέλουμε εμείς να του δώσουμε, προκειμένου να του δώσουμε τα σωστά εργαλεία. Να έχουμε τα σωστά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Οι σημερινέ κρίσει μα πρόχνουν όλου στα όρια μα. σε όρια άνευ προηγουμένου, τακτικά. Ακούσατε ποιο είναι ο κατάλογο των πέντε πιο σημαντικών ε, κατεπηγουσών καταστάσεων. L3. Έχουμε λοιπόν ε, περιπτώσεις επίπεδου 3, αλλά έχουμε και έξι κρίσεις επίπεδου 2. Είναι η Γυρία και άλλες που εξελίσσονται και ενδεχομένω να πάρουν μεγαλύτερε διαστάσει Κάθε μία από αυτές τις κρίσεις καταδεικνύει πως η αυξανόμενη κλίμακα και περιπλοκότητα των ζητημάτων απαιτεί υψηλού επίπεδου ανταπόκριση από το πρόγραμμα ψηστικής ε, βοήθειας. Γιατί δεν φτάνουν τα τρόφιμα αν δεν υπάρχει για παράδειγμα νερό, αν δεν υπάρχουν και άλλα, και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Σε 79 χώρες λοιπόν έχουμε πρόσβαση σε 80 εκατομμύρια άτομα παρέχοντας αρρωγή και τρόφιμα και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα μερίδιο μόνο των ε, ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. Αλλά έχουμε ε, παθεί και έχουμε, παρέχουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους. Ενώ παράλληλα στον, στην Παγκόσμια Οργάνωση Επιστημικής Παροχής αναπτύσσουμε και παροχή βοήθεια σε σχολεία, σε χρόνια αποστισμένα άτομα. Δίνουμε πρόσβαση σε εργασία. Και δεν το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Εταίροι μας είναι κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνδράμει μόνο οικονομικά. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας οδηγεί σε καινοτομίες, σε σημαντικά εργαλεία, προκειμένου να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο κάθε ενός δολαρίου που δαπανάτε. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ του οργανισμού μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μα δίνει καλύτερη ανθρωπιστική πρόσβαση. Ο Επίτροπο και εγώ συζητούσαμε τι προκλήσει που εμφανίζονται για να παρέχουμε βοήθεια στον κόσμο στην Ουκρανία. Πώ εξελίσσονται οι ανάγκε, πώ εξελίσσονται οι ανάγκε του λαού τη Συρίας. Αυξανόμενη επίση η απειλή του ση αλλά και των περιοχών που ελέγχονται και από την κυβέρνηση και από τους αντιφρονούντες. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στα άτομα αυτά, προκειμένου να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και να καλύψουμε τις πιο πιεστικές τους ανάγκες. Μόνο μέσω της συνεργασίας θα πετύχουμε την απαραίτητη μεταρρύθμιση που χρειάζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια και πρέπει να τα πετύχουμε αυτά. Πρέπει να πετύχουμε μεταρρύθμιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί δεν είναι γραμμικό ο χαρακτήρα των εργασιών μα. Η σχέση μεταξύ τη ανθρωπιστική αρρωγή και τη αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι γραμμικής γραμμική φύσεω. Και ο κόσμο αξίζει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην προσπάθειά μα να πετύχουμε τη μεταρρύθμιση αυτή. Το χρειάζονται αυτό και το αξίζουν. Άρα, εξ ονόματος όσους Όσον βοηθάει το πρόγραμμά μα, Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο λαό τη Ευρώπη, αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του και τη συνεχιζόμενη συνεργασία του μαζί μα. Είναι πραγματικά ανευπηγουμένου η δεσμευσή σα προ τον οργανισμό μα. Να σα ενημερώσω σε σχέση με κάποιε από τι κρίσει αυτέ που ε, πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε απερίσπαστα. το ξέσπασμα ασθενειών καταδεικνύει τι είδους προσοχή χρειάζεται η, από πλευρά του οργανισμού μας. Έχει υπηρετιστεί η εξάπλωση του εμπόλα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ε, πυρήνες ανα... αναζωπήρωσης. Χρειάζονται λοιπόν συντονισμένε δράσει ε, των κοινοτήτων, των κυβερνήσεων, των ΜΚΟ, τη διεθνού κοινότητα αλλά και του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να φτάσουμε στις μηδανικές ε, καινούργιες περιπτώσεις νόσων. Αν το κάνουμε πολύ απλά θα αναζωοποιηθεί η ασθένεια. Δεν έχει σταματήσει η κρίση επειδή έχουν ε, επιβρανδυθεί οι αριθμοί μολύνσεων. Σήμερα έχουμε, βοήθεια, έχουμε παράσχει βοήθεια σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους στους ε, επιζήσαντες, ε, στα παιδιά, στα ορφανά, σε περιοχές ε, μεγάλης μόλυνσης και έχουμε κάνει πολύ παραπάνω. Έχουμε παρέχει αεροπορικές υπηρεσίες, όχι μόνο μέσω αεροπλάνων αλλά και μέσω ελικοπτέρων για να υπάρχει πρόσβαση στους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, στα τελευταία άτομα, στα πιο απομακρυσμένα άτομα. Έχουμε δώσει βοήθεια λογιστική σε ό,τι αφορά την παροχή προστατευτικών στολών, σε ό,τι αφορά την παροχή συστήματων τηλεπικοινωνίας, η υποστήριξη πληροφορικής σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κοινότητα. Μπορείτε να μου πείτε ότι νομίζετε ότι εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα τρόφιμα. Όχι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό. Γιατί για να παρέχουμε τρόφιμα στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ του κόσμου χρειάζεται η λογιστική βοήθεια και λογιστική οργάνωση. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τι υπηρεσίε που έχουμε και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε αναπτύξει προ όφελο όλου του συστήματο ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με, με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υποστήριξη των αναγκών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Αντί λοιπόν να προσπαθούν αυτοί από μόνοι τους να αναπτύσσουν μια τεχνογνωσία που ήδη υπάρχει στους κόλπους της δικής μας οργάνωσης, τους συμπαρέχουμε εμείς τη λογιστική οργάνωση, την οργάνωση αλυσίδας παροχής τέτοιων προϊόντων. Όλη αυτή την υποστηρίξη που χρειάζεται για να μπορούν να κάνουν το έργο τους. Και αυτό είναι ένα μάθημα που μάθαμε γιατί αυτό που κάνουμε και αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε ένα οικοδόμημα που θα διασφαλίσει ότι στο μέλλον θα έχουμε αυτή τη στενή συνεργασία μεταξύ της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Παγκόσμιου Επιτιστικού Προγράμματος. Από την πρώτη ημέρα να μην συζητάμε να, για ανάπτυξη συστημάτων συνεργασίας, όχι να υπάρχουν ήδη τα συστήματα αυτά. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους διαρκούς δέσμευσης προς την Λιβυρία, Σιρελαιώνα, στην Γουινέα, η υποστήριξη της διατροφής των παιδιών και της επιστροφής στα σχολεία, της ενίσχυσης των τοπικών οικονομικών. Και ο Παγκόσμιος Επιστικός Οργανισμός κάνει σχετικές αξιολογήσεις προκειμένου να μην χάσουμε άλλη μια περίοδο σοδιάς στις χώρες αυτές. Στην Γουινέα ιδιαίτερος όπου οι αγορές εξακολουθούν να είναι δυνατές στις αγροτικές περιοχές και αρχίζουν να παρέχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράζονται τρόφιμα προκειμένου να παραμείνουν δυνατές και λειτουργικές αυτές οι αγορές και να μπορέσει να υπάρχει ελπίδα αναδόμησης των τοπικών κοινωνιών και αυτό θα επιτρέψει στους αγρότες να επιστρέψουν στη βασική τους εργασία, την δημιουργία, την παραγωγή τροφίμων. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε άμεσα σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για να συνεχίσουμε να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες υποστηρίξης και με τη δική σας διαρκή συμμετοχή και στην ε, διάσκεψη ψηλού επίπεδου για τον εμπόλα, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Και αυτό χρειάζεται, γιατί πραγματικά ο εμπόλα έχει φύγει από τα πρωτοσέλιδα και ενδεχομένω να ξαναεπιστρέψει εκεί ως η επόμενη κρίση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που το λαμβάνετε υπόψη. Στο Νότιο Σουδάν η ομάδα μας αντιμετωπίζει τεράστια εμπόδια για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια σε 3,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Παρά τις ε, μεγάλες προσπάθειές μας, οι μεταφορές μας αντιμετωπίζουν όλο μεγαλύτερες απειλές. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπα ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα και ένα αεροπλάνο κατερίφθη σχεδόν. Αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Βουλγαρία με την υποστήριξη της βουλγαρικής κυβέρνησης αλλά και άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορέσουμε να ε, εξασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πιλότων αυτών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο του πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος των ένοπλων ομάδων και πόσο δύσκολες είναι οι διαπραγματεύσεις που προαπαιτούνται προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση σε τέτοια κράτη όπου μένονται συγκρούσεις. Παρ' όλα αυτά, τώρα δρούμε για να περάσουν και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά ε, χιλιόμετρα ε, τροφίμων. Παρά λοιπόν την αυξανόμενη προβλεκότητα των κρίσεων, ό,τι περνάει από το χέρι μας το κάνουμε για να είμαστε καινοτόμοι, να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματά μας, όπως ε, η, όπως το παράδειγμα, για παράδειγμα, το πρόγραμμα για μητέρες και παιδιά. Στο Νότιο Σουδάν πέρσι, χάρη στη συνεργασία με την UNICEF, μπορέσαμε να παρέχουμε βοήθεια σε 400.000 παιδιά. Στην ε, Συρία η κρίση μπαίνει στο πέμπτο της έτος. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος καταγραμματισμός ε, της κατάστασης παροχής ε, τροφίμων. Η παροχή τροφίμων μέσω στο ιστορικό και στο εξωτερικό των ε, συνόρων και των περιοχών εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Φτάνουμε και δίνουμε βοήθεια σε 3,9 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ιστορικά εκτροπισμένοι στη χώρα μπορούν να έχουν τα τρόφιμα που χρειάζονται και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να φτάνει η βοήθεια στα άτομα αυτά. Παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσει, σε ό,τι αφορά το χαλέπι και την ενδεχόμενη πιθανότητα εκεχηρίας εκεί που θα μας επιτρέψει να έχουμε πρόσβαση στο Ανατολικό Χαλέπι για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες. Η διεθνή κοινότητα προγραμματίζει άμεση επέμβαση στις περιοχές αυτές και θα συνεχίζουμε να επεμβαίνουμε και να βοηθούμε όπου μπορούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε όλη την περιοχή, στο Λίβανο, στην Ιορδανία μέχρι και στην Τουρκία, οι πρόσφυγες παραμένουν εκτεθειμένοι, οι Σύριοι πρόσφυγες, με... εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Πέρσι, χάρη στην γρήγορη αντίδρασή σας, καταφέραμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους πρόσφυγες. Και πάλι όμως φέτος πασχίζουμε και δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των προσφύγων. Λόγω της χρηματοδότησης πρέπει να περιορίσουμε και το επίπεδο της βοήθειας που παρέχουμε. Έχουμε ήδη κάνει μείωση 30%, άρα παρέχουμε 70% της αξίας των vouchers και τώρα πρέπει να περιορίσουμε και τον αριθμό των ατόμων το προσωπικό, που θα, το, τον αριθμό των ανθρώπων που θα βοηθήσουμε. Αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους λόγω της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας που επικρατεί και στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Αν δεν παρέχουμε εμείς βοήθεια, ενδεχομένως να υπάρξει αντίκτυπο στις κυβερνήσεις αυτές, που ανησυχούν πάρα πολύ ασφαλώς ε, για το τι θα γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε περικοπή του κόστους. Όπως το σύστημα της μίας κάρτας, όπου και η UNICEF και η UNCR εξετάζει την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα της μιας κάρτας αυτής. Και επίσης ε, το πρόγραμμά μας εξακολουθεί να αποτελεί την πλατφόρμα του συστήματος αυτού. Για την Ιεμένη. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την Ιεμένη παρότι δεν είναι στα πρωτοσέλιδα σήμερα, εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εκεί τα προβλήματα 5 εκατομμυρίων ατόμων. Ξέρουμε ότι αν η πρόσβαση δεν αλλάξει, θα υπάρξει ε, εκθετική αύξηση της, προ... ανάγκης πρόσβασης στην επισητιστική βοήθεια. Άρα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες της ε, χώρας και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανασφάλεια για 10 εκατομμύρια άτομα. Σε κάποιους φτάνουμε, σε κάποιους άλλους ε, δεν μπορούμε να πάμε σε τακτικό, σε τακτική βάση. Μιλήσατε για την Ουκρανία νωρίτερα. Η... Υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσει η Εμένη σε μια κατάσταση εμπόλεμη αντίστοιχη με της Ουκρανίας. Για την Ουκρανία, η εσωτερική μετακίνηση στη χώρα και, η, και τα προβλήματα στην πρόσβαση αγοράς είναι βασικά προβλήματα ε, επισητιστικού χαρακτήρα. Η τιμή των τροφίμων στην Ανατολή έχει ε, αυξηθεί κατά 30 Έχουμε λοιπόν αυξήσει την δυνατότητά μας για να καλύψουμε τις ανάγκες εκεί. Επίσης έχουμε ε, θέσει, τοποθετήσει επισητιστική βοήθεια κοντά σε εμπόλεμες περιοχές ούτως ώστε αν επιδεινωθεί η κατάσταση να έχουμε εκεί διαθέσιμα τρόφιμα. Από τα 190.000 άτομα στα οποία δίνουμε που δίνουμε είτε χρήματα είτε ε, voucher, τους το δίνουμε για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά όταν υπάρχουν τρόφιμα. Όταν δεν υπάρχουν παρέχουμε τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν μια σύντομη εικόνα των δραστηριοτήτων μας και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε με τη βοήθειά σας για να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Ωστόσο, και παρόλες τις προσπάθειες αυτές υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες που χρειάζονται βοήθεια και θέλουν να ε, απαιτούν και, και ανάκτηση και αντοχή. Αυτό ιδίως για τις περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια και την έλλειψη πρόσβασης στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης σε θρεπτική τροφή. Όπου μπορούμε να κάνουμε δουλειά, κάνουμε για να βοηθήσουμε τις κοινότητες, τις ε, οικογένειες, τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν βιώσιμες Διαρκή λύση όταν δεν μπορούν να τη σκεφτούν οι ίδιοι. Για πολλέ από τις κοινότητε που είναι παγιδευμένες στην κρίση αυτή, είτε στι κρίσει αυτέ είτε έχουν πολιτικό χαρακτήρα ή κοινό αντίκτυπο, η δουλειά και η εμβέλεια δουλειά που κάνει το ΠΕΠ είναι αναγκαίε. Αλλά όπω είπα για πολλούς άλλου, ένα μεγάλο κομμάτι τη της ε, έγκυται στην βελτίωση τη της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας που πρέπει να γίνει όσο πιο, πιο αποτελεσματική γίνεται. Αυτό τι σημαίνει, πρέπει να υποστηρίξουμε κοινότητε με τρόπο που να είναι πραγματικές ε, πηγές αλλαγής και να στηρίζονται στην απόδοση. Στην απόδοση. Αναγνωρίζουμε ότι το να δίνουμε απλώ τρόφιμα δεν είναι αρκετό. Πρέπει, ξέρουμε ότι ο κόσμο ζητά περισσότερο από εμά και πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Να δουλεύουμε με τρόπο που θα αντιμετωπίζει, συγγνώμη, τα, προβλ... τα άμεσα προβλήματα των ατόμων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε περισσότερο ανθεκτικέ κοινότητε. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε νέε πλατφόρμε, νέα εργαλεία και σα ε, μίλησε για κάποιο. Μετρητά, βάουτσερ, ηλεκτρονικά μετρητά, τα ηλεκτρονικά βάουτσερ που παρέχουν βοήθεια και επιτρέπουν στον κόσμο να επιλέγουν τα τρόφιμα που θέλουν οι ίδιοι. Αλλά η δημιουργία πλατφορμών δίνει επίσης την ευκαιρία να έχουμε πιο αποτελεσματικό και ε, τρόπο υλοποίησης της βοήθειας αυτής. Για παράδειγμα, πέρσι στη Γάζα, το περσμένο καλοκαίρι στη Γάζα, αυξήσαμε την παροχή με βάουτσερ κατά τη διάρκεια τη ακμή τη κρίση, διπλασιάζοντα τη βοήθεια για να φτάσουμε σε 300.000 άτομα μέσα σε λίγε εβδομάδε. Αυτό μπορέσαμε να το κάνουμε διότι επενδύσαμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάτι που μα επέτρεψε να προχωρήσουμε γρήγορα. Αλλά κάναμε κι άλλα. Φτιάξαμε την πλατφόρμα, θέσαμε την πλατφόρμα μα στη διάθεση άλλων οργανώσεων που έδιναν χρήματα. και με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να αγοράσουν νερά ή υγειονομικές ανάγκες, ακόμα και ε, στολές σχολικές. Αυτό, αυτή η προσέγγιση δεν μόνο αποτελεσματική, είχε και στολε σχολικε αυτη κόστος. Βεβαίως, και μειωμενο κοστο βεβαιω εμει πρεπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και τη βελτίωση ε, τη αναγκαία ανθρωπιστική ανθρωπιστικής Ωστόσο, ταυτόχρονα πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε μια δουλειά που θα επιτρέψει να έχουμε μηδενική πείνα. Η πρόκληση που θέλουμε να πετύχουμε το 2030 όπως το έθεσε ο, είπε, ο Γενικός Δημοτές του ΟΗΕ, ζητά να μην υπάρξει κανένα ε, παιδί που να πεινάει και να υπάρχει πρόσβαση στην τροφή σε καθόλου το διάρκεια του χρόνου με ε, διπλασιασμό της παραγωγικότητας των μικρών αγροτών. Αυτό μπορεί να είναι όνειρο, είναι φαίνεται όνειρο, δεν είναι όνειρο παρά τα άνευ επίπεδα κρίσεων στον κόσμο και τον αντιτικό αντίκτυπο της αλλαγής του πληθυσμού, του κλίματος συγγνώμη, για τον πληθυσμό, πετυχάνουμε τον στόχο μας γιατί δημιουργούμε, αντιμετωπίζουμε μεθόδους βελτίωσης της, δια, διατροφής ε, με σωστές πολιτικές προς και επιτρέποντας σε όλα τα έθνη να αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση. Μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει την ώρα μου και δεν θα το πω εκτός να του θέσετε σε ερωτήσεις. Με χαρά να απαντήσω. Το να μεταφέρουμε λοιπόν από μία δυνατότητα σε μία πιθανότητα την μηδενική ποινά απαιτεί πολλούς εμπλεκόμενους πολλή προσπάθεια και μακροχρόνια, και μακροχρόνιο προγραμματισμό. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα με τη σωστή, με την καλή διακυβέρνηση. Ευτυχώς, φέτος, το 2015 είναι μια χρονιά ευκαιρία, Όχι μόνο γιατί είναι το Ευρωπαϊκό Έτο Ανάπτυξης, το είπε η Πρόεδρος, αλλά είναι και η χρονιά της οποίας, κατά την οποία μάλλον θα συμφωνήσουν τα Ηνωμένα Έθνη σε βιώσιμους στόχους ανάπτυξης και ελπίζουμε αυτή να είναι οικουμενική στόχη. Αυτό είναι μια συζήτηση μεταξύ των κρατών, διότι αφορά του πάντε στον κόσμο. Οι πάντε πρέπει να έχουν πρόσβαση σε θρεπτική τροφή ανα πάσα στιγμή προωθώντας την επένδυση, τις επενδύσεις σε δράσεις που θα πετύχουν θετικές, θετική απόδοση διατροφής, θα μπορεί να, τα κράτη-μέλη μπορεί να κάνουν το 2015 πραγματικά έτος καμπής για να τελειώσει η πείνα. Διότι φέτος μαζί με, την, με το Πεκίνο 20 και την Παγκόσμια Χρονιά Γυναίκας αποτελούν μια ευκαιρία για να για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις γυναίκες να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις ανάγκες των ιδίων αλλά και το, δυνα, δυνατότητες των κοινωνιών. Το 2015 πρέπει να είναι η χρονιά που θα διπλασιάσουμε την παραγωγικότητα των μικρών γεωργών. Το ΠΕΠΕ έχει δεσμευτεί να αγοράσει 20% όλων των ε, προϊόντων διατροφής από τους, μικρο, από τους μικρούς αγρότες. Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνεχής επένδυση στην σταθερότητα και τη μελλοντική ευημερία του κόσμου μας είναι ουσιαστική. Και η καθοδήγησή σας είναι, διότι η υποστήριξή είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι το παγκόσμιο επιστημιστικό πρόγραμμα είναι όχι μόνο ικανό, αλλά έχει και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων και να αποκαταστήσει την ζωή τους. Η επιτυχία είναι κοντά. Μαζί μπορούμε να αδράξουμε την ιστορική ευκαιρία αυτής της χρονιάς. Βεβαίως πρέπει να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να δούμε τι είναι. Ε, απλά εμπόδια στο δρόμο για τη μηδενική πείνα. Γιατί η δουλειά, το έργο του να τελειώσει, να πάψει να υπάρχει πείνα, δεν είναι έργο της επόμενης αλλά αυτής της γενεάς. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας θυμίσω τα λόγια του Νέλσον Μαντέλα όταν είπε ότι πάντα είναι φαίνεται αδύνατο μέχρι ότου γίνει. Η μηδενική πείνα μπορεί να, φαίνε, να φαίνεται αδύνατη. Και, αλλά θα είναι αδύνατη αν δεν παράσχουμε την κρατική βούληση, όπως από πλευρά σας, που θα εξασφαλίσουν ότι θα διατηρήσουμε τα, τις αναγκαίες επενδύσεις σε κονδύλια και σε ανθρώπους για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών που εξυπηρετούμε. Είτε είναι οξέα, οξύες ανάγκες, είτε μόνιμες ανάγκες. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή των ανθρώπων που εφόσον θέλουμε να πετύχουμε τη μηδενική πείνα μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήσατε θέματα, για θέματα τα οποία είναι ε, κάπως ε, καταθλιπτικά, αλλά μιλήσατε και για τις προκλήσεις και για το πώς μπορούμε να αντιπεξέλθουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε κάποιον σαν και εσάς που προσπαθεί να πιέσει, να επιτύχουμε κάτι που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Να επιτευχθεί. Είναι όμως κάτι που θα έπρεπε να είναι δυνατό, δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που να μην μπορούμε να επιτύχουμε τον 21ο αιώνα. Ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε και μερικά καλά νέα. Είπατε ότι θα μπορούσατε. Ας ακούσουμε και μερικά καλά νέα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της δουλειάς μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει ένα αποτέλεσμα, ότι κάτι είναι δυνατό, ότι έχει ξαναγίνει και ότι μπορεί να ξανασυμβεί. Ελπίζω ότι από τις ερωτήσεις θα προκύψουν κάποια καλά νέα. Επίτροπε ε, Στυλιανίδη, τέσσερις μήνες έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά που είχατε να αντιμετωπίσετε με όλες αυτές τις προκλήσεις που μόλις ακούσαμε. Ποια είναι λοιπόν η δική σας αξιολόγηση σε σχέση με το πώς πρέπει να εργαστούμε αυτή, αυτή τη χρονιά που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, ώστε να υπάρξει πραγματικά μια σημαντική αλλαγή το 2015 για θέματα τα οποία είναι πρώτης προτεραιότητας ε, στο πολιτικό θεματολόγιο. Σας δίνω το λόγο για να ακούσω τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίντα. Κυρία Εκτελεστική ε, Διευθύντρια, Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λίντα για την πρόσκλησή της ε, προκειμένου να παραστώ στη σημερινή συνεδρίαση και να ε, σας μιλήσω. Χαίρομαι όλος ε, που είμαι εδώ. Από κοινού με την Έρθαριν Κάζιν που είναι εκτελεστική διευθύντρια του Παγκοσμίου Επισητιστικού Προγράμματος δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι το Παγκόσμιο Επιθετιστικό Πρόγραμμα είναι ένας από τους βασικούς εταίρους μας στον αγώνα μας να βοηθήσουμε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ερθερίν για την ε, ε, για την εξαιρετική της ομάδα, για τους συναδέλφους τους που δουλεύουν επί τόπου, κάνουν μια εξαιρετική, καταπληκτική δουλειά βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους ε, σε μερικά από τα δυσκολότερα και πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου. Μερικές φορές μάλιστα θυσιάζουν τη ζωή τους για να σώσουν άλλους. Α, τους τιμούμε, τους χειροκροτούμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι ασφαλείς. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω εσάς, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, συγκεκριμένη Επιτροπή για την υποστήριξή σας προκειμένου να βρεθεί λύση στις περιορισμένες πιστώσεις πληρωμών για το 2014. Χάρη στη δική σας υποστήριξη αρχίσαμε αυτή τη χρονιά με ε, ισοσκελισμένες ε, υποχρεώσεις και πληρωμές. Αυτό πραγματικά είναι ένα τεράστιο βήμα και θέτει τον προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια σε στέρεα βάση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Εγώ μόλις επέστρεψα από αποστολή στο Σαχέλ, είδα από πρώτο χέρι τι θα πει ε, υποσύτηση, τι θα πει να πεινάει κανείς. Είδα παιδιά που υποσυτίζονται στο νοσοκομείο να παλεύουν για τη ζωή τους. Είδα πραγματικά την αγωνία για την επιβίωση στα μάτια των ε, μανάδων τους. Η, η κατάσταση είναι πραγματικά αφόρητη δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Είναι συλλογική μας υποχρέωση να σταματήσουμε την πείνα. Πρέπει να επιτύχουμε ε, τον στόχο της μηδενικής πείνας. Η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή αυτή καθίσταται όλο ε, και χειρότερη λόγω της έλλειψης ασφάλειας και και λόγω της πολιτικής αστάθειας. Οι μενόμενες συγκρούσεις ε, σε πολλά μέρη ε, στην περιοχή αυτή αποδυναμώνουν, υπονομεύουν κάθε προσπάθεια ε, ύπαρξης κάποιας ανθεκτικότητας και επίτευξης ανάπτυξης. Παράλληλα, δυστυχώς, το Μπόκο Χαράμ και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες αποτελούν σαφή κίνδυνο. Έχουν μια αιματηρή εκστρατεία τρομοκρατίας που αποτελεί πραγματική απειλή για ολόκληρη την περιοχή. Είναι μια απειλή την οποία δεν μπορεί να παραγνωρίζει ούτε να υποτιμά η διεθνής κοινότητα. Είχατε και μία συζήτηση με τον συναδελφο Ζων Λουί για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζετε, επισκέφθηκα την Ουκρανία πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε είδα επιτόπου τις ανάγκες. Είχα προηγουμένως επισκεφθεί τα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Μπορώ να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι αντιμετωπίζουμε άνευ ε, προηγουμένου επίπεδα ανθρωπιστικών κρίσεων, απόγνωση, αγωνία επιβίωσης, πόνο. Αυτές είναι οι λέξεις που περιγράφουν την ανθρωπιστική κατάσταση σε όλες αυτές τις περιοχές. Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε. Αυτή δυσχερής πραγματικότητα δεν πρέπει να μας σταματά. Θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές και να ελαχιστοποιηθεί ο πόνος των ευάλωτων ανθρώπων. Η συνεργασία μας με το Παγκόσμιο Επιθετιστικό Πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη. Από κοινού παρήχαμε πέρσι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια για επιθετιστική βοήθεια και τρόφιμα. Όμως αυτή η συνεργασία δεν είναι μόνο οικονομική, οικονομικής φύσεως. Είναι επίση μια συνεργασία που βασίζεται στις αρχές. Ως εταίροι πάντοτε ανταλλάσσαμε ιδέες, ε, ιδέες και ε, γνώσεις για θέματα όπως νέες προσεγγίσεις προκειμένου να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της παροχής ε, βοήθειας και σε νέες πολιτικές. Περάσαμε από κοινού από την βοήθεια με τρόφιμα στην επισητιστική βοήθεια. Χρησιμοποιούμε τους δείκτες ε, διατροφής για να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα της βοήθειας και τώρα η αντοχή είναι ε, ένα μεγάλο τμήμα της, ε, είναι ένα πλήρες τμήμα της δουλειάς μας. Συνδέουμε την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή βοήθεια και τα αντίστοιχα προγράμματα. Θέλουμε η συνδρομή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα της εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκοσμίου Επιστημιστικού Προγράμματος ε, σε, κάποια, ε, σε κάποιες από τις σοβαρότερες κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα σε κάθε μία από τις κρίσεις αυτές μέσω της ε, βοήθειάς μας, της υποστήριξής μας ε, για το, στο Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα και μέσω άλλων πολλών εταίρων ε, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Για παράδειγμα, η απάντησή μας στην κρίση της Συρίας ήταν τεράστια, μαζική. Από κοινού, με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιήσαμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή της κρίσης. Θα συνεχίσουμε βεβαίως την υποστήριξή μας ε, στο λαό της Συρίας και φέτος δεν είναι δυνατόν να χαθεί μια ολόκληρη γενεά ε, παιδιών στη Συρία. Επίσης σημειώνουμε πρόοδο στην καταπολέμηση του έμπολα. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αρχικά η διεθνής κοινότητα υποτίμησε την απειλή. Από τότε έχουμε συντονίσει καλύτερα τις ε, δράσεις μας και τώρα βλέπουμε κάποιες θετικές ενδείξεις. Όμως, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε. Δεν έχει περάσει η απειλή του έμπολα. Και όταν θα περάσει, θα πρέπει να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί να ανοικοδομήσουν την οικονομία τους, τα συστήματα περίθαλψής τους και τη ζωή τους. Η Διεθνής Διάσκεψη για την Έμπολα στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου θα συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την Έρθεριν για την συνεισφορά του Παγκοσμίου Επιστημιστικού Προγράμματος στην καταπολέμηση του έμπολα. Αμέσως ε, υπήρξαν ε, συντονιστές ε, για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε αυτές τις τεράστιες οργανωτικές προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό δείχνει πραγματικά τη δέσμευση του Παγκοσμίου Επιστημιστικού Προγράμματος και του προσωπικού του. Αγαπητοί συνάδελφοι, ανέλαβα μια δέσμευση ενώπιον της Επιτροπής σας και είμαι αποφασισμένος να κρατήσω τη δέσμευση αυτή, να τη σεβαστώ. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει τους ξεχασμένους ε, του κόσμου αυτού. Παραμένω δεσμευμένος στο στόχο να ε, βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί με μεγάλες ανάγκες, σοβαρές ανάγκες που έχουν ξεχαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν ξεχαστεί από μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Παρά το γεγονός ε, ότι ανακηρύχθηκε ως κρίση επίπεδου 3, εξακολουθεί να διατρέχει τον κίνδυνο της λύσης. Δυστυχώς. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ε, ε, βοήθειας ε, στην Κεντροαφρικανή. Παραμένουμε δεσμευμένοι να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή σε όλες τις, τις διαστάσεις. Είναι συλλογική μας ευθύνη να το πράξουμε και συλλογική μας δέσμευση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε δημιουργήσει το πρώτο, το ταμείο κατασπιστευμάτων πολλαπλών δωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε τη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση, το σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε την ε, ε, βοήθεια πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική και η απάντησή μου σε αυτό έχει τρία σκέλη. Αντοχή, διατροφή και τρόποι παροχής. Το πρώτο σκέλος, η αντοχή. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας το μακροπρόθεσμο και το, το, το βραχυπρόθεσμο και το μεσοπρόθεσμο τμήμα ε, της ε, βοήθειας όταν παρέχουμε ε, επίγουσα βοήθεια. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βοηθήσει να ε, δημιουργήσουμε αντοχή μακροπρόθεσμα και αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την επανάληψη της κρίσης. Δεύτερον, η διατροφή, η υποσύτηση εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη γιατί για το 45% των θανάτων παιδιών. Πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από υποσύτηση. Πάνω από 3 εκατομμύρια. Υποστηρίζοντας λοιπόν αυτό το σκέλος, ε, συνεισφέρουμε στη βελτίωση της αντοχής. Και επίσης συνεισφέρουμε και σε ε, μακροπρόθεσμη επισητιστική ασφάλεια των οικογενειών και των κοινοτήτων. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να μειώσει τον αριθμό των ε, παιδιών που ε, υποσυτίζονται και δεν αναπτύσσονται σωστά κατά 7 εκατομμύρια μέχρι το 2025. Όσον αφορά τώρα τους τρόπους παροχής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους οργανισμούς που προωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την μετάβαση από την παραδοσιακή επισητιστική βοήθεια στην βοήθεια ε, που συμπεριλαμβάνει ε, ρευστό και κουπόνια και όχι την παραδοσιακή αποκλειστική χρήση ε, βοήθεια της είδος, τροφίμων δηλαδή. Για να βοηθήσουμε λοιπόν την αποδοτικότητα πρέπει να αναρωτιόμαστε συνεχώ ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος παροχής όλων αυτών όλη αυτή τη βοήθεια, προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Πρέπει να αναλύουμε το πλαίσιο. Σε μερικέ περιπτώσει κατεπίγουσε, η άμεση παροχή τροφίμων είναι σημαντική. Σε μερικέ άλλε περιπτώσει ε, η χρήση των ε, κουπονιών, των vouchers είναι καλύτερη. Πρέπει πάντως αυτές οι εναλλακτικέ επιλογές να ε, αντιπαραβάλλονται πάντοτε με την επιλογή του ρευστού από την αρχή, όχι ως ε, δεύτερη ή τρίτη λύση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί το στόχο της μηδενικής πείνας μέσω των ε, προγραμμάτων μας των αναπτυξιακών. Δείτε για παράδειγμα τις βασικές μας πρωτοβουλίες όπως το Αζίρ για το Σαχέλ και το Σέρ για το κέρας της Αφρικής. Σκεφτείτε τις δεσμεύσεις μας ε, για τη διατροφή, την προσέγγιση μας για την αντοχή, την, την απάντησή μας ε, ε, στις ανθρωπιστικές κρίσεις που είναι οι τρόποι προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου της μηδενικής πείνας. μετά από την ε, σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων να πάμε μαζί να επισκεφθούμε την ε, ε, έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΠΕΠ. Είναι μια έκθεση που δείχνει σαφή παραδείγματα για το πώς αυτοί οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται επιτυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Έρφερη, ευχαριστώ πολύ Λίντα και ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή σας. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για τη δέσμευσή σα στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού ζητήματο. Και τώρα θα ανοίξω το λόγο και θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου. Τέσσερι συνάδελφοι έω τώρα έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Ντάβο Τύρ και μετά ο κύριο Γκερέρο. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερω και, τον κύριο, και την κυρία Κάζαν και τον Επιτροπό Στυλιανίδη για τα σχόλιά τους. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερος το γεγονός ότι τόνισαν ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το ξέσπασμα του έμπολα δεν έχει ακόμα σταματήσει. Να ρωτήσω τον Επίτροπο Θηλιανίδη το εξή. Ποιες είναι οι προσδοκίες από τη Σύνοδο των Βρυξελών. Δύο-τρία συγκεκριμένα αποτελέσματα που περιμένετε. Τι περιμένετε από την σύνοδο αυτή. Κυρία Κάζαν, εξηγήσατε πάρα πολύ καλά τα θέματα συνεργασίας του Παγκόσμιου Επιστηστικού Προγράμματος με άλλες οργανώσεις επιτόπου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποδομές σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η συνεργασία σας με τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων με τον ΦΑΟ και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίζετε και να πετύχετε τον στόχο της μηδενικής ανοχής στην πείνα, της μηδενικής πείνας μέχρι το 2030. Και στο τέλος αναφερθήκατε και στο στη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ καλής διακυβέρνησης και μηδενικής πείνας του στόχου αυτού. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η κατεξοχήν σύνδεση, η μοναδική σύνδεση. Το πιστεύετε κι εσείς. Ζητήσατε από τα, από τα μέλη της Επιτροπής μας να θέσουν κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις συγκεκριμένε περιπτώσεις για να μπορέσετε να απαντήσετε. Το κάνω λοιπόν. Ο κ. Γερέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο ομιλητές Σίγουρα, όταν δουλεύει κανείς με πάθος, με πεποίθηση και με συγκεκριμένους στόχους όπως ο ευγενής στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας και της πτήσης δεν υπάρχουν jet lag για τις υπερατλαντικές πτήσεις. Διαπιστώσαμε ότι η κυρία Κάουζιν με το πάθος και τη ζωτικότητά της έδειξε πως το jet lag είναι μικρό πρόβλημα, μικρό εισαγωγικό μικροαστικό αν θέλετε πρόβλημα των ε, πλούσιων τάξεων της Δύσης. Τούτου λεχθέντος υπάρχει κάτι που το βρίσκω κάπως παράδοξο και μπορεί να είναι παράδοξο για όλους. Εμείς μειώνουμε εν μέρη την πείνα στον κόσμο, ωστόσο ταυτόχρονα οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται. Σήμερα δηλαδή ως συνέπεια κάποιων επιτευγμάτων της υλοποίηση των στόχων της ηλικίας μειώσαμε τη φτώχεια, την πείνα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα η ανάγκη αντιμετώπισης επιγουσών περιπτώσεων αυξήθηκε. Έχουμε δηλαδή σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό από ποτέ ανθρωπιστικών κρίσεων μέγιστο επίπεδου. Όπως ωστόσο είπε και η κυρία Καουζίν και ο κύριος Στυλιανίδης, ε, υπάρχουν και άλλες που περιμένουν. Η Εμένη, Ουκρανία, Γάζα πάντα και άλλες τεράστιες απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βάλουμε την άμεση απάντηση, τη γρήγορη απάντηση για τις κρίσεις για τις οποίες μίλησαν οι δύο μίλητες, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να δούμε τα σχέδια και τις πρωτοβουλίες μέσω πρόθεσμα για να πετύχουμε εν ώψη του 2030 να υλοποιήσουμε την μηδενική πείνα στον κόσμο. Πιστεύω ότι με αυτή την μεσοπρόθεσμη προοπτική πρέπει να δώσουμε έμφαση στους μικρούς γεωργούς να τους υποστηρίξουμε ούτως ώστε να θέσουν τις βάσεις, να, την ρίζα για μια βιώσιμη ανθεκτική οικονομία. Σε πολιτικό επίπεδο ωστόσο πρέπει να δράσουμε για να αποφύγουμε τις αλλαγές των αγορών λόγω κλιματικών κρίσεων ή λόγω εθελούσιων ε, προβλημάτων. Εκτό βιώσαμε μια μεγάλη κρίση για τα τρόφιμα λόγω της αύξησης του τιμής πετρελαίου και την ασυνεχή σχέση μεταξύ των σημαντικότερων νομισμάτων στον κόσμο, την έλλει, της έλλειψης ε, ρύθμισης στην αγορά τροφίμων, μια σειρά δηλαδή υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων που δεν σχετίζονται με την παραγωγή των τροφίμων, αλλά σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις και τη ρύθμιση αυτών των διεθνών σχέσεων που μπορεί να έχουν εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στη φτώχεια, στη φτώχεια στον κόσμο. Όλοι ξέρουμε επιπλέον ότι σε πολλά μέρη του πλανήτη μας γίνονται μεγάλες επενδύσεις την γεωργία, στην κοινοτροφία που θα έπρεπε να μας οδηγήσουν να εξετάσουμε κατά κάποιο τρόπο για το πώς θα προτείνουμε μέτρα ούτω ώστε να είναι υπεύθυνε επενδύσεις. Να μην είναι δηλαδή επενδύσεις οι οποίες διώχνουν από την αγορά παραγωγής τροφίμων τους μικρούς γεωργούς ή να μην χρησιμοποιούν, να μην καταχρώνται των φυσικών πόρων με αρνητικό αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος που με τη σειρά του είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για πιθανές επισητιστικές κρίσεις στο μέλλον. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με την ιδέα ότι η πείνα στον κόσμο δεν πρέπει να είναι μόνο μάχη κατά της πείνας και υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων, πέραν του δικαιώματος στη ζωή βέβαια. Αποτελεί βασικό στοιχείο για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Παντού όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει ανθρωπιστική κρίση μεγάλων διαστάσεων, υπάρχει πρόβλημα έλλειψης ειρήνης, συγκρούσεων, διωγμένοι πληθυσμοί. Είναι ένα ανατροφοδοτούμενο πρόβλημα. Ο πόλεμος φέρνει πείνα, η πείνα ανατροφοδοτεί τον πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σπάσουμε κάποια στιγμή. Δύο μικρές ερωτήσεις θέλω να θέσω. Πρώτον, συμφωνώ με την ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει συμβατότητα διάφορων τρόπων παρέμβασης. Άμεση παροχή τροφίμων, κουπόνια, χρήματα, συνδυασμός των δύο. Η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει κατά πόσο είναι πιθανό να μειώσουμε την κερδοσκοπία και τη διαφθορά. Όταν αντί να δίνουμε τρόφιμα, μοιράζουμε κουπόνια, χρήματα, βάουτσερ στις εμπόλεμες περιοχές. Και πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το αρνητικό παράπλευρο αποτέλεσμα. Δεύτερον, προς τον Επίτροπο πώς θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε την επιστημιστική ασφάλεια στις πολιτικές ανθρωπιστικής βοήθειας και συνεργασίες για την ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει κάποια γενική προφανώς πολιτική για τη γεωργία, μια σειρά άλλων παραμέτρων, πώς όλες αυτές οι πολιτικές ενσωματώνονται μέσα στην πολιτική ανάπτυξη, Δηλαδή πολλές διαστάσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής θα μπορεί να έχουν επιχειρησιακό αποτέλεσμα στην επιχειρητική ασφάλεια στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε και μετά η Μαρία Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστώ την κυρία Κάζεν αλλά και τον Επίτροπό μας ε, γιατί άρχισαν τη συζήτηση με ε, σωστούς όρους με τους οποίους περιέγραψαν ε, τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Μπορεί κανείς να συνοψίσει ως εξής για όσον αφορά τα αίτια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεται σε επίπεδο παγκόσμιο ε, για την αντιμετώπιση της πείνας στον κόσμο και τις ε, φυσικές καταστροφές, την ξηρασία, ε, τους σεισμούς, τις ασθένειες που πολύ συχνά δημιουργούν προβλήματα που είναι κάποιος πιο περαστικά, μερικές φορές όμως διαρκούν περισσότερο χρονικά. Υπάρχει επίσης και μια δεύτερη κατηγορία, υπάρχουν οι αυτονομιστικές τάσεις, τέλος πάντων η ανθρώπινη βλακεία για να το πω έτσι, που όπως είπε ο Αϊνστάιν δεν έχει όρια ο Αϊνστάιν είπε ότι ο χώρος και η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια και για το χώρο δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος. Και αυτό φτάνει στο ύψιστο σημείο του όταν ε, σήμερα ε, πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σε ένα πρόβλημα ε, σε επίπεδο ε, επισητιστικό στην Ουκρανία. Ε, η περιοχή στο, στο κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται να είναι δικαιούχος ενός επισητιστικού προγράμματος. Ποιος, ποια θα είναι η λύση που θα προτείνουμε εμείς. Πάντοτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκει έναν τρόπο να ε, ε, επιβιώσει, δίνει δάνεια, μετά ε, βρίσκει έναν τρόπο να εξοφληθούν αυτά τα δάνεια, βρίσκουν βρίσκει πάντοτε έναν τρόπο να έχει ρευστό. Και εσείς πρέπει να έχετε ρευστό για να κάνετε τη δουλειά σας, Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος Και μιλάω κυρίως για τη χρηματοδότηση. Πριν από 12 χρόνια είχα ξαναπεί αυτά τα πράγματα ε, και ελπίζω ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν στην Αντίσα Μπέμπα θα είναι κάπως πιο συγκεκριμένες και θα έχουν, παρουσιάσουν περισσότερες δεσμεύσεις και θα είναι κάπως πιο αξιόπιστες από αυτά που ε, ε, ελέγχθησαν στο Μοντερέ γιατί πάρα πολλά λόγια μπορούμε να ακούσουμε, πάρα πολλές υποσχέσεις να δώσουμε που τελικά δεν θα εκπληρωθούν ποτέ και να βρεθούμε πάντοτε στην ίδια κατάσταση. Και το ερώτημά μου προς εσάς κυρίως κυρία Κάζεν, τι θα προτείνετε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα συγκεκριμένα στην Αντισαμπέμπα ε, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτές. Οι δυσκολίες αυτές ε, ανακύπτουν συνεχώς ε, και στην πρώτη κατηγορία αιτίων και στη δεύτερη που ανέφερα. Πρόκειται λοιπόν για προβλήματα διαρθρωτικά που είναι τμήμα του συστήματος τελικά. Οπότε η απάντηση πρέπει να είναι μια απάντηση σε ένα συστηματικό πρόβλημα. Οπότε το λέω αυτό για να ε, εξασφαλίσω ότι αυτή η συνάντηση στην Αντίσα Μπέμπα δεν θα γίνει μία συζήτηση ε, όπου θα αναμασάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, αλλά θα είναι μία ευκαιρία για να μιλήσουμε ειλικρινά και σοβαρά. Πείτε μας λοιπόν τι έχετε ανάγκη, συγκεκριμένα. Θέτω το ερώτημα σε εσά, αυτό όσον αφορά τώρα τον Επίτροπο, καταρχάς, αυτό που κάνετε, το κάνετε πολύ καλά και ε, φυσικά ε, νομίζω ότι ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας δεν θα το χρησιμοποιήσετε για χαζομάρες αλλά για να κάνετε πολύ καλή δουλειά. Έχετε άλλωστε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχετε την υποστήριξή μας και πραγματικά ελπίζω ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε εσά για να μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε λίγο, λίγο τα πράγματα στην αντί Σαμπέμπα γιατί πρόκειται για ένα πρόβλημα που ανακύπτει συνεχώς και η, ε, η απάντηση πρέπει να είναι αντίστοιχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μεμπρούκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Ε. Συζητάμε σήμερα προβλήματα τα οποία έχουν ε, σημαντεύσει σε όλη μου τη ζωή, όχι μόνο επειδή ήμουν από αγροτική οικογένεια και παρήγαγα τρόφιμα, αλλά επειδή ασχολήθηκα και πολύ εντατικά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάστηκα με το θέμα των, της επιστημικής ασφάλειας προ... δημοσιεύτηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση διεθνής αξιολόγηση της γνώσης, της αγροτικής γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη. Η μοναδική και κεντρική ερώτηση στην έκθεση αυτή, η οποία φτάνει τις χίλιες σελίδες και βάλε, είναι πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε την κρίση της πείνας στον κόσμο αυτό. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα και όλες οι πλευρές παρουσίασαν τη δική της άποψη. Είναι πολυδιάστατο πρόβλημα η πείνα. Ασφαλώς το ξέρουμε όλοι αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το ΠΕΠ, το Παγκόσμιο Πιστικό Πρόγραμμα, εστιάζεται εκεί που με απασχολεί και εμένα πιο πολύ, τις ε, παραγωγές, τις τοπικές, γιατί το πρόβλημα πρέπει να επιλύεται εκεί που δημιουργείται και με ιδιαίτερη χαρά άκουσα ότι αυτή είναι η βασική σας προσέγγιση. Ξέρουμε όμως επίσης ότι η πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει επιτόπου στις τοπικές κοινότητες, αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο, μορφές εμπορίου παίζουν σημαντικό ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς αντιμετωπίζουμε τη γη, ποιοι έχουν πρόσβαση στην γη, τι γίνεται, ποια είναι τα παραδοσιακά δικαιώματα αξιοποίησης των γεών. Και μεγάλο ρόλο επίσης παίζει το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα των τροφίμων, πώς υπάρχει κερδοσκοπία σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη επιρροή εδώ. Ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση από αυτά που είπατε κυρία Κάζιν. Είπατε κάθε δολάριο που επενδύεται θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί πώς θα το δαπανίσουμε για να έχει τον ανάλογο αντίκτυπο. Τι γίνεται με το πρόβλημα των φύλων από πλευρά οικονομία, ένα δολάριο που πανάτε σε μια γυναίκα τριπλασιάζεται. Το θέμα των γυναικών είναι πολύ βασικό ζήτημα όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της πείνας. Μία ερώτηση προς ε, εσάς κύριε Στυλιανίδη. Πώς μπορούμε να αναρμονιστούμε όταν μιλάμε για την παραγωγή επιτόπου και το είπατε και εσείς ότι οι μικροί αγρότες είναι αυτοί που θα πρέπει να ενισχυθούν επί τόπου, αλλά στις εμπορικές μας συμφωνίες ε, σκοπός μας είναι οι φιλελεύθερες αγορές. Ξέρουμε ακριβώς ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να προστατεύσουμε τις τοπικές αγοράς. Τι γίνεται με την απελευθέρωση του τομέα του γάλακτος στην Ευρώπη, θα υπάρξει παραπάνω παραγωγή. Υπάρχει ήδη. Και έχουμε ιδέες να στείλουμε γάλα στην Αφρική. Πώς λοιπόν μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση όσων λέμε στην εμπορική πολιτική, όσων κάνουμε στην εμπορική πολιτική και όσων κάνουμε και στην αγροτική πολιτική στην Ευρώπη και όσων γίνονται επιτόπου και των στόχων μας για την ενίσχυση των τοπικών αγορών. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο κ. Γκιόρενς είπε πριν από λίγο και ρώτησε πώς τοποθετούμαθα. Μιλήσατε για την οικονομική πτυχή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής τοποθέτηση για την πολιτική συνοχή. Και εκεί συγκαταλέγονται όλοι οι πολιτικοί τομείς. Και το εμπόριο και η αγροτική πολιτική συγκαταλέγονται. Δεν μπορούμε να προσανατολιζόμαστε για επέκταση στις παγκόσμιες αγορές σε ό,τι αφορά τη γεωργία και από την άλλη. Με εξαγωγές γαλακτοκομικών, κρέατος, να καταστρέφουμε τις αγορές. Πώς θα υπάρξει αυτή η εναρμόνιση. Um, thanks. I have a couple of questions myself. Ευχαριστώ. Και εγώ κάποιες ερωτήσεις έχω να κάνω. Κύριε Κάουζιν, δεν θα σας ρωτήσω, θα σας ρωτήσω για τα θετικά. Πείτε μας κάποιες περιπτώσεις όπου πέτυχαν τα έργα σας. Ήταν χρήσιμο να ξέρουμε περιπτώσεις. Επίσης, Μιλήσατε και οι δύο για τα βάουτσερ, τα κουπόνια. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν. Είδα μια... Είμαι ντοκιμαντέρ του BBC για το Λίβανο που έπαιρναν βάουτσερ τροφίμων στο Λίβανο. Εκεί οι ντόπιοι παραπονιόντουσαν διότι τα χρήματα ή τα τρόφιμα πληρώνονταν από το, τον ΟΗΕ και δεν ε, κέρδιζαν οι ντόπιοι φτωχοί πολίτες. Αυτά τα ζητήματα πώς τα αντιμετωπίζετε. Είναι το ίδιο πρόβλημα με το ότι οι μετανάστες έρχονται ξέρω, στη Βρετανία και μειώνουν, οδηγούν σε μείωση των ε, μισθών. Πώς χειρίζεστε την κατάσταση, έχετε κάνει ανάλυση και προς τον Επίτροπο τώρα. Αναφερθήκατε, είπατε ότι βραχυπρόθεσμη ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να, έχει, να έχουμε στο μυαλό μας και το μακροπρόθεσμο. Στην, πριν ήρθατε μιλούσαμε για την Ουκρανία και κάποιοι από την υπερτερμοστία του ΟΗΕ τους πρόσφυγες μας είπαν ότι κάποια κράτη-μέλη δεν συντονίζουν την βοήθεια με άλλες χώρες που παρέχουν βοήθεια ε, και πάνε, στέλνουν τη, βοήθεια με κοντέινερ που το ΟΗΕ θεωρεί ότι δεν είναι καλό εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό μέσα στην Ένωση πριν ξεκινήσει να παρέχεται η βοήθεια. Το, κάναμε, το είδαμε με τον έμπολα. Μπορούμε να έχουμε μια αντίστοιχη προσέγγιση για τον προπολογισμό τώρα. Να πω χαίρομαι που βλέπω ότι το πρόβλημα του προπολογισμού λύθηκε αυτό το πρόβλημα και όλοι οι επιτροποί θέλουν να συνεργαστούμε μαζί του χρόνου τόσο ώστε να ξεκινήσουμε νωρί τη δουλειά το 2016, να μην αρχίσουμε τις ίδιε μάχε κάθε χρόνο. Ίσως θα έπρεπε αυτό να το ξεκινήσουμε νωρίτερα, μην επανέλθουμε δηλαδή μόνο τον Οκτώβριο για να μπαίνουμε στις ίδιε συγκρούσει για τον προπολογισμό. Αυτά. Η κυρία Κάζιν καταρχάς. begin with the um, questions from... Πολλές ερωτήσεις από τον κύριο Στήρ. Είχατε πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, πώς η συνεργασία μας για τη μείωση της, για την επιτευξη της μηδενικής ε, πείνας με το ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι πολύ σημαντικός οργανισμός. Εμείς ε, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τους μικρούς αγρότες, η παραγωγικότητα και την παραγωγικότητα της υποστηρίζοντας ότι θα έχουν τα σωστά εργαλεία. Η εμπειρία εκεί είναι στο ΦΑΟ, όχι σε εμά. Δουλεύουμε από κοινού λοιπόν για να εξασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τα σωστά εργαλεία, τους σωστούς σπόρους, τους γεωργούς. Και ότι ε, για να επενδύσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μετά, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την πρόσβαση στην αγορά, αγοράζοντας από τους μικρούς γεωργούς, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ξέρουν πού μπορούν να πουλήσουν τα, τα, τα τρόφιμά τους και πού μπορούν να πάρουν καλύτερες τιμές. Επίσης, συνεργαζόμαστε για την οικοδόμηση εντοχής. Ποιες ευκαιρίες δηλαδή υπάρχουν για να δώσουμε νέα εργαλεία στις κοινότητες που μπορεί να εντοπιστούν από τον ΦΑΟ και εμείς να δουλέψουμε με ΜΚΟ και ντόπιε οργανώσεις για την υλοποίησή τους χρησιμοποιώντας τρόφιμα ή μετρητά για να υποστηρίξουμε αυτό που λέμε food for asset development ή food for work δηλαδή δημιουργώντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Έτσι δουλεύουμε όχι μόνο τόπου αλλά και σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Π.χ. δουλέψαμε για την, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ήταν από κοινού δουλειά, παρέχοντας πληροφορίες ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σαν στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ελπίζουμε να το συνεχίσουμε. Για την ορθή διακυβέρνηση. Η σωστή διακυβέρνηση είναι κλειδί, συμφωνώ. Όταν μιλάμε για οξύες ανάγκες. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε οξύες ανάγκες γιατί δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση. Όταν όμως λέμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες διαρκείς λύσεις που θα επιτρέψουν τη διατήρηση της αντοχής του πληθυσμού, του resilience πρέπει να υπάρξει εμπλοκή των κυβερνήσεων. Αυτό δεν είναι δουλειά του ΠΕΠ αλλά του UNDP, άλλων οργανώσεων που δουλεύουν με τις οργανώσεις για την διαμόρφωση του σωστού πλαισίου πολιτικής που θα υποστηρίξουν θέματα ορθής διακυβέρνησης. Και αυτό είναι ο λόγος τον οποίο ε, δουλεύουμε μαζί για να πετύχουμε αποτελέσματα ανάπτυξης. Και εσείς και οι και οι πρόεδρος με ζήτησαν για καλές ιστορίες εμείς δεν σκεφτόμαστε συχνά την Κορέα ως χώρα που χρειαζόταν επισητιστική βοήθεια. Αλλά παλιά ήταν βασικοί ε, δέκτες επισητιστικής βοήθειας, αλλά υπήρξε σωστή διακυβέρνηση, βελτιώθηκε η εκπαίδευση και έτσι η χώρα αυτή είναι πλέον δωρητής. Μια άλλη χώρα που δεν σκεφτόμαστε συχνά σήμερα ήταν η Κίνα η Κίνα ήταν η χώρα που πριν από 15 χρόνια δίναμε τα περισσότερα, την περισσότερη επιστημιστική βοήθεια. Πιστεύω ότι ποτέ δεν καταφέρει να φάει, να, να, να τρέφεται μόνη της. Είδατε που πήγε η Κίνα. Γουατεμάλα πριν από λίγο καιρό. Είχα πάει στη Γουατεμάλα και μιλούσα σε γυναίκες γεωργούς. Μια γυναίκα μου είπε τους είπα τι, τι σημαίνει ότι εσείς τώρα έχετε δυνατότητα όχι μόνο να καλλιεργείτε τρόφιμα για να τρώτε αλλά για να πουλάτε και τα τρόφιμα στην αγορά και να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας. μου απάντησε αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ ο άντρας μου. Έμεινε εδώ. Μιλάμε λοιπόν για θέματα που δημιουργούν ικανότητες, δυνατότητες στις κοινότητες. Αυτό σημαίνει επενδύουμε για το μέλλον. Μια πρόσφατη περίπτωση είναι η Ουγγάντα, πιο πρόσφατη. Εμείς εκεί δουλεύουμε για να υποστηρίξουμε όχι μόνο την διαμόρφωση αντοχής αλλά και την μείωση των απολειών μετά τη συγκομιδή. Στην υποσαχαρική Αφρική 40% της συγκομιδής χάνεται σε κακή, με κακούς, από κακούς χειρισμούς. Έχουμε ένα πρόγραμμα πέρυσι, ξεκινήσαμε μάλλον, που οδήγησε σε 80% μείωση των απολειών μετά τη συγκομιδή. Η Παγκοσμία Τράπεζα επενδύει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 100.000 αγρότες στην Ουγκάντα να μειώσουν τις απώλειες αυτές. Να προγράμματα που αλλάζουν την κατάσταση. Για το θέμα, το ερώτημα που έφεσε ο κ. Γκέρενς, την κερδοσκοπία και τη διαφθορά και τον αντίκτυπο που έχει κάτι τέτοιο στα τρόφιμα και αν είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε βάουτσερ η πραγματικότητα είναι ότι οι πολιτικοί δεν θέλουν να μπουν, δεν θέλουν να μπω σαν πολιτικό στα θέματα κερδοσκοπίας και διαφθοράς, αλλά αυτό που είδαμε από το 2008 και μετά οδήγησε όχι μόνο σε κερδοσκοπικές δράσεις και αύξηση των τροφίμων, αλλά και είδαμε και το πώς αντέδρασαν οι χώρες, ιδίως ε, στις, στις απαγορεύσεις εξαγωγής και τον, ε, την επίπτωση που είχαν στις χώρες εισαγωγών, που ήταν φτωχές χώρες κυρίως και δεν είχαν, ε, δεν είχαν να μην είχαν πρόσβαση σε τρόφιμα και εδώ εξοδήγησαν σε εξεγέρσεις τροφίμων που θυμόμαστε. Το να έχουμε κουπόνια αντί για μετρητά δεν θα άλλασε την κατάσταση. Εμείς τι προτείνουμε για την Αντίσα τρία πράγματα. Ένα, μεγαλύτερη πολιετή ευέλικτη χρηματοδότηση που μας επιτρέπει να επενδύουμε σε προγράμματα που δίνουν αποτελέσματα και όχι μόνο εκροές. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να μελτρήσουμε τα αποτελέσματα και ελπίζουμε οι δωρητές να μας δώσουν την ευελιξία που θα επιτρέψει να έχουμε αυτή τη μακρό πρόθεσμη προσέγγιση. Δεύτερον, καινοτόμα χρηματοδότηση για εκροές. Το Food Secure, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα υποστήριξης το, και χρηματοδότησης που θα επιτρέπει επενδύσεις των δωρητών με ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μπορεί το World Food Program να διατηρήσει την υποστήριξή του σε πληθυσμούς μεταξύ κρίσεων. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Έχεις μια κρίση. Επενδύεις στην οικοδόμηση εντοχής, πιστεύουμε στο διπλό δρόμο, χρηματοδοτούμε, μετά καταστα... καταλαγιάζει και μετά μέχρι την επόμενη κρίση ε, σταματάει η χρηματοδότηση και ξαναπέφτει πίσω ο πληθυσμός. Οι δραστηριότητε οικοδόμηση αντοχή, όπω και οι δράσει τι οποίε επενδύει η Ένωση στην περιοχή του Σαχέλ, επιτρέπουν υποστήριξη καινοτόμων έργων που παρέχουν τη δυνατότητα σε γυναίκες για παράδειγμα να ε, αυξήσουν τις αντοχές τους πολλώντας λαχανικά για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της περίοδου των βροχών. Όταν έρθει όμως η επόμενη κρίση ο αριθμός των ανθρώπων που υφίστανται αντίκτυπο θα ήταν μικρότερος αν, από ό,τι στην προηγούμενη κρίση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δίνουμε μόνιμη βοήθεια που επιτρέπεται από την ευέλικτη χρηματοδότηση. Μόνο έτσι θα αλλάξουν οι εκροές. Ή, θα αλλάξουν συγγνώμη τα αποτελέσματα. Άλλη λύση θα ήταν να ζητήσουμε από τις χώρες να επενδύουν στην δική τους τις δικές του αστηριότητες επιστημιστικής ασφάλειας και διατροφής. Η εκτελεστική, το εκτελεστικό γραφείο του ΠΕΠ μας έδωσε εξουσία να παρεμβαίνουμε στις μεσαίου εισοδήματος χώρες μόνο αν πληρώνουν οι χώρες αυτές για το έργο του ΠΕΠ. Αυτό πρέπει να είναι μια δέσμευση που προκύπτει από την, θα προκύψει από την αντίσταση Αμπέμπα όταν περισσότερες χώρες θα, θα επενδύουν και θα ξέρουν κατά πόσον αυτό μπορεί να γίνει σε πολυμερές επίπεδο για την υποστήριξη των δράσεων αυτών. Τέλος, πρόσβαση στη γη και κερδοσκοπία στα τρόφιμα. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο δουλεύει πάλι το ΦΑΟ. Τον υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε τι διαφορέ δραστηριότητε της αλλά είναι ένας τομέα που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο. Τώρα η υποστήριξη, μάλλον τα κουπόνια. Τα κουπόνια δουλεύουν, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη σωστή δουλειά για να αξιολογούμε κατά πόσον τα βάουτσερ ή τα κουπόνια βοηθούν τις κοινότητες. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες αγορές, να υπάρχουν ισχυρές αρκετά στιβαρές αγορές και να μην δίνουμε βάουτσερ ή μετρητά σε μια κοινότητα που θα οδηγήσουν μετά σε πληθωρισμό και να Έχουμε κόσμο που μπορεί σήμερα να μην χρειάζεται βοήθειά μας, αλλά να αυξηθούν οι τιμές και να χρειαστεί τη βοήθειά μας στο μέλλον. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που με τη γενναιοδότητα τους μας βοηθάμε. Εμείς αναλύουμε τις αγορές για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε πληθωριστικές τάσεις σε περιοχές όπου δουλεύαμε πάντα όχι μόνο για να προστατεύσουμε αλλά και να βελτιώσουμε για την ερώτηση του κατά πόσον δεν επηρεάζουν τα μέσα εισοδήματα, τα, κουπό, τα κουπόνια μέσα εισοδήματα στις περιοχές αυτές μειώνοντας έμεσα τους μισθούς. Εμείς πρέπει να κάνουμε στοχοθετημένη δράση δίνοντας βοήθεια μόνο σε όσους την έχουν ανάγκη. Αν δεν θες να δουλέψεις, α, μάλλον αν δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να παίρνεις ε, βοήθεια, διεθνή βοήθεια. Στην Ιορδανία, για παράδειγμα, αυτοί που παίρνουν βοήθεια δεν επιτρέπει να δουλεύουν. Αν δηλαδή κάποιο παίρνει χρήματα ή ε, βοήθεια από εμά, δεν πρέπει να μπορεί να δουλεύει. Η ικανότητά τους δηλαδή ε, για να διατρέφουν την οικογένεια παραμένει, αλλά δεν φύγεται η, η, η κοινότητα υποδοχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπος, έχει το λόγο. Τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου για το Mother Tank. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε στο τέλος η Έρθαριν, επειδή το έζησα on the ground στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Η Λίντα έθεσε ένα θέμα, το οποίο έχει απόλυτο δίκιο πολλές φορές ο τρόπος που παρέχεται η βοήθεια δημιουργεί κάποια προβλήματα στα θέματα της αγοράς εργασίας στη συγκεκριμένη χώρα. Και αυτό είναι πολύ έκθυλο στο Λίβανο. Έχει επηρεαστεί η αγορά εργασίας και είναι ολοφάνερο. Ε, όμως στην κοιλάδα Μπεκά, κάτι σε σχέση που είπε και η Έρθαρη, βρήκα μια οικογένεια, η μάνα με έξι παιδιά, σε ένα μικρό δωμάτιο που τους παρήχαμε εμείς ως διεθνείς δωρητές, έπαιρνα μια βοήθεια, αλλά υπήρχε και ένα παιδί, ο μεγάλος γιος, στα 16 του, που έπρεπε να δουλεύει για να μπορέσει να φτάνει σε ένα επίπεδο επιβίωσης στην οικογένεια. Ειλικρινά επειδή θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και είναι διαφορετικά να βλέπεις τα θέματα από το γραφείο σου και διαφορετικά να τα βλέπεις on the ground. Θέλει εξαιρετική εξειδίκευση για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό να είμαστε ειλικρινεί. Το σύστημα πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα έχει ατέλειες. Αλλιώς θα, είμαστε, θα εθεροπαντούμε. Λοιπόν, ο στόχος ποιος είναι. Αυτές οι ατέλειες να είναι οι λιγότερες δυνατές. Αυτή είναι η αξία. Και έχω την εντύπωση τουλάχιστον από τη μικρή μου εμπειρία επί του εδάφους on the ground ότι υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα να βρίσκει τρόπους να περιορίζει αυτές τις ατέλειες. Μπαίνω και σε μια άλλη ερώτηση η οποία τέθηκε από τον κύριο Γκέρενς τον οποίο ευχαριστώ για τα καλά λόγια για το θέμα του corruption, της διαφθοράς. Είναι ένα μεγάλο στίχημα να περιορίσουμε όσο μπορούμε το ενδεχόμενο corruption. Και νομίζω ότι σε αυτό το χώρο υπάρχει μια δυνατότητα συνεχούς βελτίωση. Δεν υπάρχει αφιβολία. Νομίζω το παραδέχεται και η Ότι έχουμε δυνατότητα συνεχούς βελτίωση. Αυτό όμω που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς θα γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των χρημάτων. Και είναι ένα μεγάλο στίχημα στο θέμα του να φέρουμε σε ίση μοίρα τα commitments με τα, με τα payments. Χρειαζόμαστε, ναι, πιο αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων. Χρειαζόμαστε καλύτερο accountability. Και είναι ενδεχομένως ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε και στην Κωνσταντινούπολη στο International Conference το οποίο είναι από τα κύρια ζητήματα μαζί με την καινοτομία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο από την αρχή κάποιες από τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση του συνάδελφου του Ενρίκη. Καταρχήν, συμφωνώ απολύτως ότι ναι, ενώ περιορίζεται το θέμα του υποσυντισμού, εν αυξάνονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες οι έκτακτες ειδικά. Η ανατροφοδότηση όπως πολύ σωστά είπες έχει σχέση με πολιτική πραγματικότητα. Ξεκινά από το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικοί λόγοι. Είναι γι' αυτό που λέμε δυστυχώς οι ανθρωπιστικά προβλήματα χρειάζονται πολιτικές λύσεις. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συζητούσαμε πριν με την Ερθράδιν, για το Σουδάν. Είναι αδιανόητο σήμερα δύο άνθρωποι στο Σουδάν να δημιουργούν αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Και να τους παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα αδύναμη να βρει λύση άμεσα. Είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου δημιουργεί άμεσο πρόβλημα. Νιώθω πάρα πολύ άβολα μέχρι και ντροπή αυτό το γεγονός. Ότι δεν βρήκαμε λύση σε μια κατάσταση στο Σουδάν η οποία οφείλεται ουσιαστικά σε δύο προσωπικότητες οι οποίες έχουν φέρει την κατάσταση εκεί που την έχουν φέρει. Ο Ντίβορ με ρώτησε για τα expectations, για τις προσδοκίες από το, για το Ebola Conference. ήδη από τον κατάλογο των όσων έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν φαίνεται ότι θα είναι μια εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή και κατά την προσωπική μου άποψη το πλέον σημαντικό είναι ότι θα έχουμε εάν δεν συμβεί κάτι την παρουσία και των τριών ηγετών των τριών affected countries Λιβερίας, Σιέρα Λεόνε και Γουινέας. Θεωρώ ότι εκτός του ότι θα συζητήσουμε σοβαρά προβλήματα για την επόμενη μέρα, όπως είναι το healthcare system, το rebuild του healthcare system, θα μπορούμε με τέτοιο επίπεδο συμμετοχής προέδρων κυρίως να συζητήσουμε regional cooperation. Τουλάχιστον on the ground αυτό που αντιλήφθηκα και το μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε στην αρχή της διάδοσης του ιού προερχόταν από την αδυναμία στο κρίσιμο red point των τριών συνόρων, των χωρών των τριών συνόρων δεν υπήρχε αυτό το στοιχειώδες regional cooperation. Προσωπικά όπως είδα την κατάσταση on the ground θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αυτή την, το regional cooperation στο πιο ψηλό επίπεδο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε νέες κρίσεις και ενδεχομένως νέα φαινόμενα είτε από μαλάρια είτε από χολέρα. Το άλλο που θα συζητηθεί είναι αυτό που υπενόησε πολύ σωστά η Έρθαλη ότι ναι, χρειαζόμαστε αποκατάσταση του καβερνας. Και αυτό που συνέβηκε παραδείγματο χάρη στην Κορέα και φτάσαμε σήμερα να είναι δωρητή, ουσιαστικά είναι το ότι αποκαταστάθηκε το καβερνας. Το μεγάλο πρόβλημα και στις τρεις αυτές χώρες ξεκινάει ίσως και από το καβερνας. Γι' αυτό θα συζητηθεί και έχω την μεγάλη προσδοκία ότι όλα αυτά μαζί βέβαια με συγκεκριμένες προτάσεις για το healthcare system, για τα θέματα ανάπτυξης, θα είναι ουσιαστικές συζητήσεις που θα δημιουργήσουν τη νέα αρχή για την περιοχή. Βέβαια, δεν υποτιμώ, δεν αγνοώ καθόλου το γεγονός ότι η περιοχή έχει ήδη εκδηλώσει προβλήματα Ασφάλεια που προέρχονται από την Πόκο Χαράμ και από τις εξελίξεις στο βόρειο Μάλι. Είδα στον ΚΑΟ, ήμουν πριν δύο μέρες και αντιλήφθηκα επακριβώς το τη σύνδεση του insecurity με όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ανθρωπιστική κρίση και την ανάπτυξη. Δυστυχώς πρέπει και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει το comprehensive approach. Το χρειαζόμαστε, τουλάχιστον το δικό μας Relex Committee γίνονται μεγάλες συζητήσεις με βάση την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Yes. Νομίζω πολλά ήδη έχει απαντήσει και είμαστε στην ίδια γραμμή με την Έρθαρη να συμφωνήσω απολύτως με την Μάρια για το θέμα ότι χρειάζεται να στηρίξουμε την τοπική παραγωγή και θεωρώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα θέματα του πορτοφολίου μου χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως το Αζίρ στο Σαχέλ και το Σέαρ στο χώρο ΦΑΦΡΙΚΑ αυτό επιδιώκουν. Και δεν νομίζω να επηρεάζεται από οποιαδήποτε άσκηση άλλης πολιτικής αυτή τη στιγμή τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να συμβαίνει σε άλλες περιοχές. Και κάτι τελευταίο για το, θέμα του budget συμφωνώ απολύτω με τη Λίντα. Πρέπει να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Να πω κάτι τελευταίο για το θέμα του cash and voucher και, και τη βοήθεια σε είδος. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όμως πιστεύω ότι εξαρτάται απολύτως από τις συνθήκε στην κάθε διαφορετική χώρα. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και να επιλέγεται κατά χώρα, κατά περίπτωση η καλύτερη και η πιο αποτελεσματική διαδικασία. Αλλού το cash and voucher, αλλού η, βοήθεια σε είδους. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε είμαι στην Επιτροπή αυτή, απολαμβάνω τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Well, can I thank both our speakers for... Να ευχαριστήσω και του δύο ομιλητέ που μα παρουσίασαν με τέτοιο καλό τρόπο τι μεγάλε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στο μέλλον και να σα καλέσω παρακαλώ όλους σας να έλθετε στην ε, φωτογραφική έκθεση στον τρίτο όροφο Family Meal. Θα ανοίξουμε λοιπόν την έκθεση αυτή. Θα γενιάσουμε την έκθεση και θα προσπαθήσουμε να επιστήσουμε την προσοχή του Κοινοβουλίου ολόκληρου στα θέματα που αντιμετωπίσουμε αύριο. Θα λέμε αύριο στις 10.45 και πρώτα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Στις 9 λοιπόν για τους συντονιστές και στις 10.45 για τους υπόλοιπους. Και ευγενικά η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλό απόγευμα.